Good morning, Καλημέρα σας. Ξεκινώ την δεύτερη, τη συνεδρίαση της δεύτερης μέρας της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Στην ημερήσια διάταξη έχουμε την κοινή συνεδρίαση με την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ανταλλαγή απόψεων με τον Γιέρζη Πομιανόφσκι, ο οποίος είναι εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Πρικοδότησης της Δημοκρατίας και θα παρουσιάσει την πρώτη ετήσια έκθεση του Ιδρύματος αυτού. Για τον κύριο Πομιανόφσκι θα ήθελα να κάνω μια σύντομη εισαγωγή. Πρωτού γίνει εκτελεστικός διευθυντής του Ιδρύματος, ήταν αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών στην Πολωνία, στην κυβέρνηση του κύριου Τούσκ. Αυτό ήταν ήδη και στη δεκαετία του πριν τη δεκαετία του 80 ήταν από τους ακτιβιστές της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στην Πολωνία όταν ήταν φοιτητή. Αργότερα υπήρξε δημόσιος υπάλληλος στο Υπουργείο Παιδείας. Μετά υπεύθυνο για τα θέματα Αφρικής και Μέσης Ανατολής στο Υπουργείο Εξωτερικών, πρέσβης στην Ιαπωνία, εργάστηκε στα θέματα συνεργασίας με το πρόγραμμα ανάπτυξης των Ηνωμένων Πολιτειών, προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης και συνεργασίας επίσης αντιμετώπιση συγκρούσεων και φυσικών καταστροφών και ήταν από το 2006 μέχρι το 2008 υπεύθυνο για το πρόγραμμα ανάπτυξης της Πολωνίας και συνεργασίας. Ο στόχος σημερινής συζήτησης είναι να ε, πάρουμε τις πληροφορίες σε σχέση να πάρουν πληροφορίες για το ρόλο του Ιδρύματος για τη Δημοκρατία, του Endowment for Democracy, που υποστηρίχθηκε ιδιαίτερα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπήρξε και μια πρωτοβουλία της Πολωνίας για την προώθηση της δημοκρατίας, εκεί όπου δεν έχει ακόμα αποκτήσει στέρεες ρίζες, επί τη βάση της πρόσφατης εμπειρίας και της Πολωνίας. Το Ίδρυμα αυτό λοιπόν είναι μια κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, και των, ιδρυμάτων, των ε, Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων. Είναι ένας ανεξάρτητος φορέας που υπόκειται στον βελγικό ρόλο. Έχει έτσι μια ευελιξία που του επιτρέπει να δώσει με ταχύτητα χρηματοδότηση μέσα σε λίγες μονάχα και να δράσει σε χώρους όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει δυσκολίες να δράσει λόγω των διαδικασιών που συνάπτονται με το δημοσιονομικό κανονισμό η γεωγραφική εστίαση του Ιδρύματος για τη Δημοκρατία είναι οι, κυρίως οι γειτονικέ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες και από την έποψη αυτή ο κύριος Πομιανόφσκι είναι σε πολύ καλή θέση να λάβει υπόψη <clears throat> τις προτεραιότητες για την υποστήριξη πρωτοβουλειών για την κοινωνία των πολιτών και την ενίσχυση της δημοκρατίας και στην ανατολική μας γειτονιά αλλά και στην νότια γειτονιά μας. Και έτσι θα ακούσετε από τα χείλη του με ποιο τρόπο χρησιμοποιούνται τα κονδύλια τα οποία δόθηκαν στο Ίδρυμα για τη Δημοκρατία, πώς έχουν κατανεμηθεί σε μια σειρά σχεδίων και στα ε, βορειοανατολικά και στα νότια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω το ότι οι συνάδελφοί μας στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ιδίω ο Αντζέι Τζιμπ, ο οποίος είναι από την Πολωνία. Μπορούν να μας δώσουν περισσότερα στοιχεία και μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια έκθεση πρωτοβουλίας για το Ίδρυμα για τη Δημοκρατία. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στον κύριο Πομιανόφσκι. Ευχαριστώ Πρόεδρε και μέλη της Επιτροπής που επιτρέπεται στο Ταμείο μας να κάνει την πρώτη του ετήσια έκθεση. Επίσης καθήκον μου είναι να κάνω αυτή την ετήσια, να αυτή την ετήσια έκθεση. Αρχίζω εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη μας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ΕΠΕΞ και όλους τους κοινοβουλευτικούς γιατί χωρίς την υποστήριξή σας θα αντιμετωπίζαμε πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες. Σε κάθε φάση της προπαρασκευαστικής διαδικασίας της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Δημοκρατία μας βοηθούσατε και μπορέσατε να απομακρύνετε και μερικά γραφειοκρατι... μερικούς γραφειοκρατικούς και πολιτικούς φραγμούς. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικός ο ρόλος του Κοινοβουλίου και φαίνεται και στις διοικητικές δομές μας. Ο Έλμαρ Μπροκ είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Αλεξάνδρ Λάντσδορφ της Εκτελεστικής Επιτροπής. Εννέα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνολικά είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και προέρχονται από 8 διαφορετικές χώρες. Νομίζω ότι είμαστε πολύ ιδιαίτεροι οντότης. Έχετε μπροστά σας, ελπίζω, ένα αντίτυπο της έκθεσής μας και θα σας αναφέρω ορισμένες από τις κύριες ιδέες της. Η απόφαση για την ίδρυση του ΦΕΝΤΕΜΗ, του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Δημοκρατία, έχει, είχε γίνει για να αντιμετωπίσει ορισμένα νέα στοιχεία στο γεωπολιτικό παιχνίδι και σήμερα είμαστε πολύ πιο πολιτικά ευαίσθητοι γιατί η ίδρυσή μας σηματοδοτεί νέες τάσεις και στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία από, κεντρο, από κρατοκεντρική προσέγγιση σε πιο αποκεντρωμένη με όλη την κοινωνία των εταίρων να συμμετέχει και την κοινωνία των πολιτών στην κάθε χώρα αυτή. Το ΕΙΔΑ έχει σε λιγότερο από τρεις μήνες από τότε που άρχισε τον Ιούλιο του 2013 να λειτουργεί πλήρως όπως προβλεπόταν. Πάνω από 1200 αιτήματα για στήριξη βοβλήθηκαν και 120 δωρεές χορηγήθηκαν μέχρι σήμερα. Εξισορροπημένες μεταξύ ανατολικών και νότιων χωρών της πολιτικής γειτονίας. Στη σελίδα 19 τα λέμε αυτά. Ο αριθμός των ετοιμάτων που μας υποβάλλονται είναι κυρίως από τις ανατολικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά τα πιο υψηλά, οι πιο υψηλές δωρεές χορηγούνται στις νότιες ώρες. Αυτό είναι ενδιαφέρον φαινόμενο. Το ΕΙΔ υποστηρίζει τον πολιτικό ακτιβισμό ή δραστηριότητες που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν με τα παραδοσιακά χρηματοδοτικά όργανα χρηματοδοτεί οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών και που υποστηρίζουν την ειρήνη και τη δημοκρατία. Αυτά τα λέει στη σελίδα 12. Μερικά παραδείγματα. Πολλοί έχουν λάβει δωρεές από το ΕΕΔ, από τους ακτιβιτές του Μαϊντάν μεταξύ των οποίων μερικοί είναι αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες όπως και η Σβετλάνα Ζαλιτσούκ. που τώρα έχει γίνει, ευρωβουλευτής έχει γίνει στην Ουκρανία και υποσχέθηκε να συνεχίσει να πιέζει για τις μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι ένα μόνο παράδειγμα από τις επιτυχείς δραστηριότητες μας χρηματοδότησης δραστηριοτήτων. Γενικά, συνολικά, το ΕΕΔ έχει χορηγήσει 6,5 εκατομμύρια δωρεές από 2.000 μέχρι 200.000 η καθεμία και υποστήριξε δραστηριότητες ακόμα και σε πολύ δύσκολες πολιτικές συνθήκες και συνθήκες ασφαλείας. Από τη σελίδα 9 της έκθεσής μας τα λέει αυτά. Τα πιο ευαίσθητα ή λεπτά προγράμματα δεν τα αναφέρουμε γιατί για αυτά υπάρχει ειδική διαδικασία που λέγεται Beneficiary Protection Procedure για να μην βγουν αυτά πέρα από τη γραμματεία. Είπα και πριν ότι βασιζόμαστε κυρίως σε την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία στις 15 χώρες που συμπεριλαμβάνει αυτή. Τον πρώτο χρόνο δεν θα σας εκπλήξει αν μάθετε ότι ασχοληθήκαμε κυρίως με τις χώρες που, που αντιμετώπιζαν μεγάλες δημοκρατικές προκλήσεις καθώς και εμείς. Στην Αίγυπτο και το Αζερβαϊζάν οι προκλήσεις αυτές ήταν και είναι σχετιζόμενες με τον συνδιακώς μειωνόμενο χώρο της ελευθερίας. Στο Αζερβαϊζάν διάφορες δωρεές, αυτή ε, ε, αυτοί που έλαβαν δωρεές Πολλοί από αυτούς είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή και πάγωσαν οι λογαριασμοί τους. Γιατί θεωρήθηκε ύποπτη η συνδρομή από το εξωτερικό και υπήρχε όλο και περισσότερη παρενόχληση από την αστυνομία. Η πρόσφατη τροπολογία ή αλλαγή του ποινικού δικαίου στην Αίγυπτο και αυτή που προτείνεται στο Αζερβαϊζάν θα καταστήσει κάθε έμβασμα από το εξωτερικό παράνομο στη Συρία δημοκρατικά κινήματα ειρηνικά χρειάστηκε να λειτουργήσουν σε πολύ εχθρικό περιβάλλον και έχουν καταντήσει όμοιροι και του καθεστώτος και των ακραίων δυνάμεων. Το Ταμείο πάντως το Ίδρυμα αναγνωρίζεται διεθνώς ως χρήσιμο γιατί δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο δημοκρατικός χώρος και η στήριξη των ε, δραστηριοτήτων της κοινωνίας των πολιτών συνεχώς μειώνεται. Οι κυβερνήσεις θα πανούν λιγότερα για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα, προγράμματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Νομίζουμε λοιπόν ότι καλύπτουμε ένα κενό που είναι τελείως απαραίτητο σε μια εποχή όπου χρειάζεται ένωση δυνάμεων. Εμείς συνεργαζόμαστε με όλους τους διεθνείς προμηθευτές δωρεών για τη δημοκρατία και στην Ευρώπη και διατλαντικός. Υπάρχουν γερμανικά πολιτικά ιδρύματα, ολλανδικά, το NDI, IRI, NED, Freedom House, German Marshall, Euro-Mediterranean Foundation και πολλά άλλα ιδρύματα και think tanks δεξαμενές σκέψεις δηλαδή που βασίζονται πολλά στις Βρυξέλλες. Η υποβοήθηση και στήριξη της δημοκρατίας είναι σημαντική. Τα γεωπολιτικά παιχνίδια βέβαια απαιτούν όλο και περισσότερη στήριξη των, της δημοκρατίας αλλά υπάρχει και το θέμα της σταθεροποίησης και ασφάλειας που αποτελεί πολλές φορές μια δικαιολογία για να μειωθούν οι δημοκρατικές ελευθερίες. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν όλο και ισχυρότερη πίεση να αποδείξουμε τη χρησιμότητά μας και αυτό είναι θεμητό. Στην πράξη όμως αυτό συχνά σημαίνει ότι αναγκαζόμαστε να τονίζουμε κυρίως τα βράχη πρόθεσμα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε και όχι τα υπόλοιπα ενώ κανονικά χρειάζεται πολύς χρόνος για να μπορέσει κανείς να πει ότι έχει στηριχθεί η δημοκρατία και έχει αυξηθεί ο δημοκρατικός χώρος. Άρα όσοι θέλουν να βοηθήσουν τη δημοκρατία πρέπει να επιλέξουν. Χρειάζεται πιο σοβαρή αντιμετώπιση και πιο μακροπρόθεσμη ή ελαφρύτερη όπως προγράμματα σε μερικές χώρες που θα μπορούσαν να παγώσουν για να μην εκτεθούν οι ακτιβιστές τους σε, να υποκύψουν σε πιέσεις από τις κυβερνήσεις. Σόφρον επιλογή όμως είναι αυτή ή όχι. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφαρμόσουμε την ίδια προσέγγιση σε κάθε περιβάλλον. Αντίθετα, θα πρέπει να αναπτύξουμε νέε καινοτόμε στρατηγικέ για να έχουμε ένα πιο καλό τρόπο αντιμετώπιση. Πρέπει να εξασφαλίσουμε επίση τη σωστή χρηματοδότηση και την βελτιστοδοξία του Ιδρύματό μα. Με τον τρόπο αυτό, χάρη στι εθελοντικέ συνεισφορέ των κρατών μελών και του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να εξασφαλίσουμε τον πυρήνα της χρηματοδότησης και αυτό ήταν και η βασική σύλληψη του Ιδρύματος. Για να μπορούμε να αποφέρουμε καρπούς θα πρέπει να έχουμε τους απαραίτητους πόρους. Και, Ευρωπαϊ... και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο να ασκήσουν πίεση στις κυβερνήσεις των κρατών μελών για να συμβάλλουν ιδιαίτερα στο πρόγραμμα αυτό. πρέπει να πω ότι η χρηματοδότηση δεν είναι ο μόνος τρόπος για να υποστηρίξουμε τη δημοκρατία. Πρέπει να συνεχίσουμε τη διπλωματική πίεση στα κατασταλτικά καθεστώτα για να εξασφαλίσουμε ότι οι ακτιβιστέ δεν θα είναι θύματα καταστολής. Πιστεύω ότι με το να ξαναστρέψουμε τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα κοινωνικό στροφό παράδειγμα, όπως είδαμε στην Τινησία, την Αίγυπτο και την Ουκρανία, είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τον επιθετικό πουτινισμό και άλλες ιδεολογίες οι οποίες στρέφονται κατά της δημοκρατίας και των δημοκρατικών θεσμών και μειώνουν τον χώρο της κοινωνίας των πολιτών και των δημοκρατικών δικαιωμάτων. ένα ορατό κομμάτι αυτής της εργασίας θα συνεχίσει να γίνεται από το Ίδρυμα για τη Δημοκρατία και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε οποιοδήποτε ερώτημα έχετε σε σχέση με την έκθεσή μας. Ευχαριστώ. Thank uh, Πραγματικά ήταν μια παρουσίαση πλήρης. Σας ευχαριστώ για την έκθεσή σας. Δεν ξέρω τώρα αν οι συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο. Ανδρέη Τσίπ, Πρέντα μετά, Μπούτι Κόφερ και Γκόμες. Έχουμε 40-45 λεπτά ακόμα για τη συζήτηση αυτή. Παρακαλώ να μην τα ξεπεράσουμε και να είστε μετρημένοι στο χρόνο που χρησιμοποιείτε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πιωμανός, και συγγνώμη για την εξαιρετική πράγματι παρουσίαση την οποία μας έκανε μόλις. Ε, αυτά τα οποία είπατε σήμερα είναι πάρα πολύ χρήσιμα και τα εκτιμώ δεόντως. Σας ευχαριστώ επίσης και για το έγγραφο το οποίο ε, μας ε, δώσατε. Ενάμιση χρόνο δουλεύετε, αλλά τα αποτελέσματα υπάρχουν ήδη. Η πρωτοβουλία σας είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη. Να θυμηθούμε τη βάση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Βασιστήκαμε στην εμπειρία της λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης, όπως επίσης και στα πλαίσια της ε, συμφωνίας και της εταιρικής συνεργασίας ε, με την Μεσογειακή Λεκάνη. προσπαθήσαμε να βάλουμε στο, στο κέντρο των σχέσεών μας με όλη αυτή την περιοχή και τις χώρες αυτές ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα μέσα που είχαμε στη διάθεσή μας ε, ήταν με επαρκή ε, σχετικά αλλά δεν ήταν σε θέση να κινητοποιηθούν ταχύτατα διότι τα προβλήματα απαιτούν άμεση παρέμβαση από πλευράς μας. Το άμεσο βέβαια δεν σημαίνει και πρόχειρο πόσο μάλλον λανθασμένο ή στρεβλό. Τέθηκαν πολλές, πολλά αιτήματα για χρηματοδοτήσεις, άνω των χιλίων αιτήσεων κατετέθησαν και αυτό και μόνο δείχνει την αναγκαιότητα του συγκεκριμένου αυτού μέσου. Φυσικά και δεν στάθηκε δυνατό να χρηματοδοτήσουμε όλους όσους το ζητούσαν, γιατί τελικά μόνο 150 αιτήσει ελήφθησαν υπόψη και έτυχαν ε, της επιθυμητής χρηματοδότησης. Αυτά όλα δείχνουν όμως ότι ε, είναι σημαντικός ο ρόλος ε, της συγκεκριμένης δομής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξ αρχής υποστήριξε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Υπήρξε μια τροπολογία στην έκθεση De Kaiser η οποία ασχολήθηκε με τα θέματα του εκδημοκρατισμού. Αυτό έγινε και μάλιστα στην αρχή της Πολωνικής Προεδρίας πριν λίγα χρόνια. και αμέσως, μετά την, αμέσως πριν μάλλον την αρχή της Πολωνικής Προεδρίας ο Υπουργός Στανόφσκι είχε καταθέσει τις προτάσεις του στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τότε. Μας είχε εξηγήσει τις βασικές αρχές λειτουργίας του συγκεκριμένου μέσου. Ένα μέσο το οποίο θα έπρεπε να είναι πιο ευέλικτο από τα ήδη υπάρχοντα τότε, ένα μέσο πιο διαδραστικό και πιο ταχύ στις δυνατότητες παρέμβασης που είχε, το θέμα δεν ήταν απλά να βοηθήσουμε κάποια πολιτικά ιδρύματα ή κάποιους πολιτικούς οργανισμούς, αλλά και την ίδια την κοινωνία των πολιτών. Και μάλιστα στα πλαίσια της πολιτικής άνοιξης ε, δεν υπήρχε ε, δημοκρατικός θεσμός τον οποίο να χρηματοδοτήσουμε. Ήταν λοιπόν πιο περίπλοκα τα πράγματα και γι' αυτό τέσσερα έγγραφα επηρέασαν άμεσα την δημιουργία της συγκεκριμένου ε, μέσου. Η έκθεση The Kaiser, η ετήσια έκθεση για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Αυτά ε, είναι το 2012 και τα δύο. Ο κύριος Χάουιτ ήταν μάλιστα εισηγητής και ο κύριος Χάουιτ είχε πει ότι θα πρέπει να αναφερθούμε στην έκθεση αυτή ε, και στην υποστήριξη που θα δώσουμε για την δημιουργία του Ιδρύματος ε, ή του Ταμείου αν θέλετε για την Δημοκρατία. Ακολούθησε η έκθεση Ταβάρες στις 29 Μαρτίου του 12. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε το κείμενο το ιδρυτικό του μέσου αυτού και ε, συζήτησε με το Συμβούλιο τις συνθήκες δημιουργίας του συγκεκριμένου νέου μέσου. Η έκθεση η σχετική ε, την εισήγαγε ο κύριος Λάμστορφ. Εδώ προστίθεται το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από πλευράς του ε, δέχτηκε τις τροπολογίες του Συμβουλίου σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης ε, για την περίοδο 2014-2020, την επόμενη δηλαδή προγραμματική. Και αυτό μας επέτρεψε να βρούμε ε, μαζί με το Συμβούλιο κάποιες λύσεις για την χρηματοδότηση που προσδίδουν περαιτέρω νομική σταθερότητα και ε, ασφάλεια στην λειτουργία του συγκεκριμένου Ιδρύματος. Όπως είπε ο κύριος Πομιανόφσκι, οι κυβερνήσεις μειώνουν τις άμεσες ε, επιχορηγήσεις τους στη στήριξη των δημοκρατικών θεσμών και ε, καλύπτεται το κενό από τα νέα μέσα, μεταξύ των οποίων το δικό μας αυτό μέσο για τη δημοκρατία. Αυτό λοιπόν απέδειξε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα στα διάφορα κράτη-μέλη και μπορεί να δώσει κίνητρα στα κρατημέλη έτσι ώστε να βοηθήσουν ε, για τον εκδημοκρατισμό. Ήδη 13 φορές μέλη υποστηρίζουν την ε, πρωτοβουλία και έχει εγγραφεί μάλιστα και η Ελβετία. Αυτό που έχει σημασία εδώ είναι ότι αυτού του είδους ε, η αποτελεσματική και μακροπρόθεσμη βοήθεια οικονομική ε, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από μια κάποια διάρκεια στον χρόνο. Και γι' αυτό ακριβώς προσπαθήσαμε να επιλέξουμε το σωστό πλαίσιο λειτουργίας της. Ε, υπογραμμίσατε κύριε Πομιανόφσκι τα θέματα που άπτονται της αποτελεσματικότητας του μέσου όπως επίσης και της εικόνας του μέσου προς το κοινό. Από τη φύση του το μέσο σε ορισμένες χώρες η επέμβασή του δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερος ορατή και ο καρπός των εργασιών του ε, θα γίνει γνωστός και αντιληπτός μετά από κάποια χρονική περίοδο. Καταλαβαίνω βέβαια ότι αυτοί οι οποίοι χρηματοδοτούν συγκεκριμένα τα κράτη-μέλη θα επιθυμούσαν τα αποτελέσματα να είναι ορατά άμεσα και όχι να επενδύουν σε δραστηριότητες οι οποίες θα αποδώσουν σε υστερότερο χρόνο. Όμως και αυτές είναι απαραίτητες και θα τις εξετάσουμε όταν κληθούμε πλέον να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα και την λειτουργία του νέου αυτού μέσου. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η γεωγραφική εντολή ή η γεωγραφική κάλυψη. Ασχολείται με 13 χώρες μέχρι σήμερα το συγκεκριμένο αυτό μέσο, γειτονικές όλες άμεσα, αλλά υπάρχουν βέβαια ανάγκες και σε άλλες γεωγραφικές περιφέρειες. Είναι ένα δίλημα το οποίο έχουμε μπροστά μας. Στην παρούσα φάση δεν έχει νόημα να αναζητήσουμε τη διεύρυνση της γεωγραφικής κάλυψης, διότι οι οικονομικές μας δυνατότητες είναι περιορισμένες. Είναι όμως τίθεται το θέμα της πιθανής στο μέλλον τουλάχιστον αύξησης της γεωγραφικής εμβέλειας του συγκεκριμένου μέσου. Υπάρχουν πολλές χώρες ε, όμορες ε, στις οποίες η δραστηριότητα του Ταμείου και του είναι πάρα πολύ δύσκολη και να μην πω ανέφικτη. Να σας αναφέρω μόνο το παράδειγμα της Συρίας. Αναφερθήκατε και εσείς κύριε Πομιανόφσκι στα της Συρίας. Στην χώρα αυτή υπάρχουν οι εξτρεμιστές από τη μία, οι δυνάμεις του καθεστώτος από την άλλη και οι δύο αυτές δυνάμεις είναι εχθρικές στην δραστηριότητα και στην λειτουργία του ε, μέσου το οποίο έχουμε πλέον στη διάθεσή μας. Αυτό ήταν ένα παράδειγμα. Λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία θα ανταλάβουμε ε, υπόψη μας στα πλαίσια της αξιολόγησης την οποία θα κληθούμε να κάνουμε από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τζιμ. Ε, Και τώρα ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πομιανεύσκη. Ε, σας ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίασή σας. Λαμβάνω τώρα τον λόγο εξ του ΕΛΚ αλλά και ως νέο μέλος του του Διοικητικού Συμβουλίου του EED, όπως ελέγχθηκε προηγουμένως. Έχουμε προτείνει να εκπονήσουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας για το Ίδρυμα για τη Δημοκρατία και είμαι σίγουρος ότι εμείς θα συνεργαστούμε πολύ στενά για να εξασφαλίσουμε ότι η έκθεση αυτή θα μπορέσει να ενισχύσει τις δραστηριότητες του Ιδρύματος για τη Δημοκρατία. Θέλω να σας συγχαρώ λοιπόν για την εκκίνηση με τόσο αποτελεσματικό τρόπο του προγράμματος αυτού. Βλέπω ότι όλα λειτουργούν πολύ καλά και υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες οι οποίες έχουν λάβει χώρα. Υπήρξε σημαντική υποστήριξη από την έκθεσή σας. Με εντυπωσιάζει ο αριθμό των δραστηριοτήτων που έχει αναπτύξει το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία. Θέλω να θέσω τώρα ορισμένα ερωτήματα σε εσά. Καταρχήν για κάτι το οποίο λέτε στην έκθεσή σας. Λέτε ότι παρά το γεγονός ότι είναι εύκαμπτη διαδικασία σε ό,τι αφορά την κατανομή των πόρων εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία. Αποτελεί αυτό απλώς μια μορφή αυτοκριτικής ή υπάρχει και η δυνατότητα να ευκαμπτοποιήσετε ακόμα περισσότερο τις διαδικασίες σας. Βλέπω πίσω ότι υπάρχουν τρεις χώρες για τις οποίες υπάρχει ιδιαίτερη στόχευση του Ιδρύματος και για τις οποίες όμως δεν έχετε <clears throat> καταφέρει να παρουσιάσετε τις δραστηριότητές σας. Στην Συρία είναι πολύ φανερό ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει κάτι, αλλά μεταξύ αυτών των χωρών είναι και η Αλγερία. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πολιτικά εμπόδια ή απλώς συνέβη ότι δεν μπορούσατε να παρουσιάσετε τις δραστηριότητες του, του Ταμείου σας στην Αλγερία. Τέλος. Δεν θα σας ρωτήσω κατά πόσο είναι δυνατόν σε ένα ορατό μέλλον, σε ένα βραχυπρόθεσμο μέλλον, να καλύψετε και περισσότερες χώρες. Αυτό έχει ήδη προταθεί φυσικά. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο από τον Ιούνιο μέχρι τώρα υπήρξαν ε, και κάποιες ε, προσπάθειες να συμπεριληφθούν και περισσότερες χώρες στο πρόγραμμά σας. η ομάδα μου σίγουρα είναι έτοιμη να υποστηρίξει τη δράση του Ιδρύματος για τη Δημοκρατία και ιδίως σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων. Και το ΕΛΚ είναι απόλυτα δεσμευμένο προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέω. Ευχαριστώ, Κρίστιαν. Αλλάζω λιγάκι τη σειρά των ομιλητών. για να ακολουθούμε τις πολιτικές ομάδες. Για τους σοσιαλιστές ο κύριος Παντσέρη, ο οποίος είναι και ο συντονιστής των. Ευχαριστώ τον κύριο Πομιανόσκη για την παρουσία του εδώ και την παρέμβασή του. Θα συμφωνήσει μαζί μου ότι εμείς ε, βιώνουμε μια ε, ιστορική φάση κάπως ιδιαίτερη και αμφισβητούνται οι γεωπολιτικές αναφορές βλέπουμε ότι αυξάνονται οι σειράξεις στον κόσμο και αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά η, δυνα... ανάγκη παρέμβασης για την πρόθεση της δημοκρατίας, κάτι που δυστυχώς όμως συμβαδίζει και με την έλλειψη οικονομικών πόρων. Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω κάποιες σκέψεις και για τις δραστηριότητες τις οποίες μέχρι τώρα έχει διεξάγει το Ίδρυμά σας τέσσερα σημεία. Νομίζω ότι είναι και οι τέσσερις στόχοι του ε, Ιδρύματος αυτού. Ο πρώτος στόχος αναφέρθηκε και από τους δύο προλαλήσαντες. Θα πρέπει ακριβώς να έχουμε ένα βλέμμα εντελώς ανοιχτό, 360 μοίρες. Δεν θα πρέπει να περιορίσουμε την προσοχή μας σε συγκεκριμένες μόνον χώρες. Δεύτερον, Κατανοώ αυτά τα οποία είπατε και οι δύο, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε μια ισορροπία ανάμεσα στην Ανατολή της Ευρώπης και τον Νότο. Το λέω αυτό γιατί έχει ξεκινήσει η συζήτηση και στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχουν υπάρξει πολιτικές αντιπαραθέσεις σχετικά με το αν θα έπρεπε να προκρίνουμε τις σχέσεις μας με την Ανατολική Ευρώπη είναι μια πρόταση την οποία εν μέρη καταλαβαίνω, αλλά έχουμε όμως σοβαρά προβλήματα και στο Νότο. Δεν μπορούμε να τα αγνοούμε. Ένα τρίτο στοιχείο είναι μια ερώτηση την οποία θα ήθελα να σας θέτω. Μιλάμε για μια δυνατότητα παρέμβασης η οποία βασίζεται σε προτεραιότητες στρατηγικής φύσεως. Θα πρέπει βέβαια ακριβώς επειδή συγκεντρώνουμε την προσοχή μας και επιλέγουμε προτεραιότητες θα πρέπει να δείξουμε τα αποτελέσματα της κατά παρέμβασής μας στην και ευρωπαϊκή κοινή γνώμη για να ενδιαφερθεί για το πρόβλημα. Ξέρουμε το τι γίνεται τελευταία στη Μέση Ανατολή, βλέπουμε τα προβλήματα που δημιουργεί το καλυφάτο όπως λέγεται και βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη για παρεμβάσεις σε αυτό τον τομέα και σε επίπεδο πολιτιστικό, όχι μόνο πολιτικό, για την πρόθεση της δημοκρατίας. Και τέλος, τελευταίο σημείο, συνέργειες με άλλα όργανα, έτσι ώστε να αποφύγουμε τις επικαλύψεις των μεμονωμένων δραστηριοτήτων. Θα ήθελα τη γνώμη σας επ' αυτού. Σας ευχαριστώ κύριε Παντσέρη. Η κυρία Φώτιγκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Πομιαπτόφ. Θα ήθελα να σας ε, ευχηθώ κάθε επιτυχία στο έργο σας και φυσικά θα ήθελα να συνεχίσω εκεί που σταμάτησε ο προλαλή σα για τι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ χαίρομαι για το γεγονό ότι ένα Πολωνό, ο οποίο είναι επικεφαλή του Ιδρύματο αυτού, το οποίο έχει σαν στόχο να μεριμνήσει για όλες τις ανάγκες παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα ευρύ γεωγραφικό χώρο. Αυτός ο χώρος φυσικά έχει δημιουργηθεί και μετά την Αραβική Άνοιξη. Αυτό κατεδεικνύει ότι οι κοινωνίες και τα κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης έχουν τη δυνατότητα να δεσμευτούν για να μεταλαμπαδεύσουν την εμπειρία τους στις χώρες αυτές που αντιμετωπίζουν προκλήσεις και δυσκολίες σε ό,τι αφορά την εγκαθίδρυση και την εδραίωση της δημοκρατίας. Θα ήθελα να τονίσω ότι στη συζήτηση αυτή θα ήθελα να μην υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ γεωγραφικών περιοχών. Θα πρέπει να μπορέσουμε να δούμε ποιες είναι οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και όχι από ποιο γεωγραφικό χώρο προέρχονται. Έχουμε λοιπόν προκλήσεις και στα νότια και στα ανατολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως δεν πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε μία μονάχα περιοχή. Είναι υποχρέωσή μας να αντιμετωπίσουμε με τον κατάλληλο τρόπο όλες αυτές τις προκλήσεις. Γι' αυτό πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση μεταξύ μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Ο κύριος, Τσου, ο κύριος Λάμστορφ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Πομιανόφσκι για την παρουσίαση που μας έκανε. Θέλω να πω τώρα τα εξής. Προφανώς πρέπει να ευχαριστήσω καταρχήν τον Διευθυντή και τους συνεργάτες του στο Ίδρυμα αυτό για το Ταμείο αυτό, για το Ίδρυμα για τη Δημοκρατία. Όταν τότε είχαμε διαπραγματευτεί με το Συμβούλιο για το Ίδρυμα αυτό, υπήρχαν ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία θέλανε να έχουν μια πολύ μικρή γραμματεία. Αλλά βλέπετε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό αιτήσεων και είναι απαραίτητο να υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση και επαρκής στελέχωση για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το Ίδρυμα αυτό όλες τις αιτήσει. Δεύτερο, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν ε, συνεργαστεί με το Ταμείο αυτό στο Διοικητικό Συμβούλιο και εδώ θέλω να αναφέρω συναδέλφους που δεν είναι παρόντες όπως ήταν ο Ινάσιος Αλαφράγκα, η Βερονίκ Ντεκεζέρ κτλ. Στο παρελθόν οι νέοι τώρα συνάδελφοι οι οποίοι θα προέλθουν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ταμείο αυτό έχουν μια εμπειρία ήδη στην δραστηριότητα αυτού του ταμείου και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε καλύτερες κοινέ πρωτοβουλίες μεταξύ της Κομισιόν, της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης των Κατών Μελών και φυσικά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πολύ καλό το ότι εκπροσωπείται και η Κομισιόν και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Έχουμε λοιπόν μια ιδιαίτερη δομή, ένα ιδιαίτερο σχήμα με το οποίο μπορούμε να λειτουργήσουμε. Και τρίτον θέλω να ε, ευχαριστήσω και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Γιατί έχουμε όχι μονάχα βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εννέα βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και τρεις από την κοινωνία των πολιτών, οι οποίοι συμμετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή. Πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν μεγάλη εμπειρία από την ίδια τους την προσπάθεια να προωθήσουν τους στόχους της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες τους και έχουν μπορέσει να λειτουργήσουν σε ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες και πιστεύω ότι και οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, όπως και οι εκπρόσωποι των κρατών μελών, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την εμπειρία των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών για να γίνει πιο αποτελεσματικό και επιτυχές το σχέδιο και το πρόγραμμα του Ιδρύματος. Θέλω και αυτού λοιπόν του εκπροσώπου τη κοινωνία των πολιτών να του ευχαριστήσω. Ποιε είναι τώρα οι προκλήσει που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε τρει κύριε προκλήσει που πρέπει να τι αντιμετωπίσουμε ω Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα, αυτό το οποίο ονόμασα pushback, το λεγόμενο κύμα απόθεσης και περιστολής όλων των διεκδικήσεων που έχουν να κάνουν με τη δημοκρατία, το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα για τα ιδρύματα για τη δημοκρατία, τα γερμανικά, τα ολλανδικά και άλλα, τα οποία υφίστανται μεγάλες πιέσεις από τα αυταρχικά καθεστώτα. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν είναι πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την προσπάθεια να περιοριστεί η δράση όλων αυτών των ιδρυμάτων τα οποία θέλουν να υποστηρίξουν τις οικουμενικές αρχές και ελευθερίες. Ένα δεύτερο θέμα, και εδώ στρέφομαι περισσότερο προς τους συναδέλφους από τις χώρες όπου μπορεί να υπάρξει καλύτερη λειτουργία, είναι το θέμα της χρηματοδότησης. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος και για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Ο κύριος Παντσέρη είχε εδώ απόλυτο δίκιο όταν είπε ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και την ε, γεωγραφική ισορροπία μεταξύ Ανατολικής Ευρώπης και Νότιας γειτονιάς της Ευρώπης Αλλά βλέπω ότι χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία δεν έχουν συνεισφέρει ακόμα στο Ταμείο. Χαίρομαι για το γεγονός ότι η Ισπανία είναι έτοιμη να χρηματοδοτήσει, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά οικονομικά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά η Ισπανία είναι έτοιμη να συνεισφέρει στο Ταμείο αυτό. Θα ήθελα να ελπίζω ότι οι συνάδελφοί μας από τις χώρες όπου δεν έχει γίνει ακόμα καμιά έχει υπάρξει χρηματοδότηση του Ταμείου θα ασκήσουν πίεση για να μπορέσει να υπάρξει και μια θετικότερη στάση των χωρών της σε, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση αυτή. Τέλος, όπως είπε και ο κύριος ε, Γκριμπς, πρέπει να έχουμε υπομονή για το έργο αυτό. Η υποστήριξη της δημοκρατίας δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει μηχανιστικά. Δεν είναι ότι περνάμε ορισμένα σχέδια και προγράμματα και με αυτόν τον τρόπο ξαφνικά δημιουργείται ένα δημοκρατικό κλίμα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολλές προκλήσεις, πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα, γι' αυτό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα το Ταμείο αυτό να λειτουργεί και σε χώρους οι οποίοι δεν είναι οι συμβατικοί, οι συνηθισμένοι χώροι εργασίας ενός τέτοιου ιδρύματος. Και τέλος, μία ε, πρόκληση που ευτυχώς δεν υπάρχει πια, είναι το να δημιουργήσουμε εδώ στις Βρυξέλλες μια συνένεση μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων σε σχέση με το νόημα και την αναγκαιότητα ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία και έχουμε ήδη μια θετική στάση από την Κομισιόν, την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και το Συμβούλιο και φυσικά είναι φανερό ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει ε, πλήρως αυτήν την ε, αυτό το εγχείρημα. Έχουμε περάσει λοιπόν την φάση της ε, διαπραγμάτευσης για τη λειτουργία του Ιδρύματος και χάρη σε αυτή τη συνένεση περνάμε λοιπόν σε μια φάση εφαρμογής του προγραμματός του και θέλω να ευχαριστώ στον κ. Πομιανόφσκι και τους συναδέλφους του κάθε επιτυχία και ελπίζω ότι θα ξεπεράσουμε τις ε, γεωγραφικές τους γεωγραφικούς περιορισμούς και θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο τη δραστηριότητα αυτού του Ιδρύματος και θα έχουμε τους απαραίτητους πόρους και εύχομαι κάθε επιτυχία στις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λάμστοφ. Είναι φανερό ότι ορισμένοι από εμά έχουν μια ιδιαίτερη ε, υποχρέωση να κάνουν τα απαραίτητα για να εξασφαλίσουν τον προϋπολογισμό. Η κυρία Λόζινγκ έχει τώρα το λόγο. Ε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ε, παρουσίαση και μετά από αυτά που ελέγχθηκαν και από τους συναδέλφους θέλω να πω ότι το εργαλείο αυτό έχει δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Από τη μία πλευρά υπάρχει μια πολυπλοκότητα που πρέπει να αντιμετωπίσετε. Από την άλλη πλευρά όμως είναι απαραίτητο να υπάρχει μια οκίτητα στον τρόπο με τον οποίο αντιδρά το Ταμείο. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα του ελέγχου και της διαφάνειας που δεν πρέπει όσο και δύσκολο να είναι να παραμεληθούν. Γι' αυτό θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα για τον έλεγχο του προϋπολογισμού των μέσων του Ταμείου αυτού. Βάσει του άρθρου 10 του καταστατικού σας, έχει την δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί εν μέρη ή πλήρως από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην έκθεσή σας λέτε ότι το Ίδρυμα αυτό υπόκειται στο βελγικό δίκαιο σε ό,τι αφορά την, τον οικονομικό έλεγχο. Θα ήθελα να ξέρω στο μέλλον αν μπορούν να υπάρχουν βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 4 του καταστατικού να υπάρχει έλεγχος από τρίτους φορείς, δηλαδή από εξωτερικούς λογιστικούς ελέγχους, αν θα μπορούσε να γίνεται αυτή, αυτός ο έλεγχος για τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Και επίση έχω ένα ερώτημα σε σχέση με τις ΣΕΝΤΟΥ. Λέτε στο προήμιο της έκθεσής σας ότι η υποστήριξη της δημοκρατίας έχει ξαναγυρίσει στη γεωπολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως ο ρόλος του Ιδρύματος αυτού είναι πολύ πιο σημαντικός πια. Επίσης αναφέρεται κάπου αλλού ότι ο... για κάποιο διάστημα η δράση της υποστήριξης δημοκρατίας είχε παραμεληθεί σε κάποιο βαθμό και εκεί αναφέρεται την... το ρόλο του Ιδρύματος αυτού. Στο άρθρο 2 Παράφως ε, παράγραφος 2 λέτε ότι μεταξύ άλλων οι αναδιόμενοι ηγέτες θα πρέπει στις χώρες όπου υποστηρίζει το Ταμείο Δημοκρατία θα πρέπει να υποστηριχθούν. Δεν ξέρω τι ακριβώς όμως σημαίνει αυτό και με ποιο τρόπο πώς μπορούν μη κυβερνητικοί οργανισμοί και οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών και αναδυόμενοι ηγέτες όπως λέτε μέσα εισαγωγικά με ποιο τρόπο μπορούν να εντοπίζονται σε ένα τόσο πολύπλοκο πλαίσιο όπως αναφέρατε που δρά το Ταμείο θα ήθελα να ξέρω πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Σκεφτείτε την Αίγυπτο, σκεφτείτε την ε, Ουκρανία. Πώς μπορεί κανείς να επιλέξει και επιβάσει ποιων κριτηρίων θα γίνεται αυτή η υποστήριξη των αναδυομένων ηγετών στις χώρες αυτές. Και έχω και ένα συγκεκριμένο ερώτημα για την Ουκρανία, η οποία αντιμετωπίζεται σαν συνολική ε, οντότητα. Υπάρχουν και περιφερειακές ε, διαφοροποίησεις που γίνονται και υπάρχουν και δραστηριότητες οι οποίες αφορούν τις ανατολικές και νοτιοανατολικές περιοχές σε ό,τι αφορά τους αναδυόμενους ηγέτες ή τις ΜΚΟ Ποιε ακριβώ δραστηριότητε υποστηρίζονται εκεί. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον Διευθυντή Πομιανόσκη για την παρουσίασή του. Να τον ευχαριστήσω και αυτόν και το προσωπικό της υπηρεσίας του για τη δουλειά την οποία ολοκλήρωσαν τον πρώτο χρόνο εκφράζουμε την ικανοποίησή μας γιατί βλέπουμε ότι ε, πλέον αποκτά μορφή μετά από ένα χρόνο ε, μόνον λειτουργίας πιο συγκεκριμένη και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και να συνεργαζόμεθα με το ε, Ίδρυμα αυτό. Συμφωνώ μαζί σας και Πομιανόφσκι ότι η κατάσταση συνεχίζει να είναι πάρα πολύ οξυμένη στο γεωγραφικό χώρο με τον οποίο ασχολείστε. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, μεταξύ των οποίων και το δικό σας, για να στηρίξουμε τους πρωταγωνιστές της δημοκρατικής αλλαγής. Θα συμφωνήσω επίσης μαζί σας κύριε και όπως είπατε και στην εισαγωγή σας ότι κάποιες σκέψεις βραχυπρόθεσμες στον τομέα της ασφάλειας και της σταθεροποίησης δεν θα πρέπει να μας αποτρέπουν να δούμε γενικότερα το πρόβλημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έρχομαι τώρα σε συγκεκριμένα σημεία. Αναφερθήκατε ειδικά στην κατάσταση στην Αίγυπτο και μιλήσατε για το πόσο δύσκολη γίνεται σιγά σιγά η κατάσταση στην Αίγυπτο. Μπορείτε παρακαλώ να μας πείτε ε, τους τρόπους της, ε, δυνα, της, τις δυνατότητες που έχετε για παρέμβαση που να βελτιώσει την κατάσταση στην Αίγυπτο. Δεύτερον, η στήριξη αυτών που δεν την χάνουν στήριξη από πουθενά. Από την άλλη βέβαια βλέπουμε ότι μία μειοψηφία ομάδων που ζητούν βοήθεια πράγματι ε, βοηθούνται τι μπορεί να γίνει στο μέλλον έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις δυνατότητες παρέμβασής μας και ποσοτικά. Κάποιοι άλλοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στην λεγόμενη γεωγραφική εντολή, εμβέλεια, κάλυψη, ό,τι επιθυμείτε. Θα ήθελα να προσπαθήσουμε να είμαστε ο λίγων προ, προβλεπτικοί προς την κατεύθυνση αυτή να μην χρησιμοποιούμε μονίμως σαν καραμέλα το επιχείρημα της έλλειψης πιστώσεων. Να σκεφτούμε ότι αν πράγματι έχουμε να αντιμετωπίσουμε με χαίνοντα προβλήματα σε μια ευρύτερη γεωγραφικά περιοχή, τότε μπορούμε να ζητήσουμε επιπλέον πιστώσεις. Σαν παράδειγμα, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και την ρωσική δημοκρατία στις χώρες με τις οποίες ε, ασχολούμεθα. Τώρα για τις οικονομικές ε, συνεισφορές ε, των διαφόρων χωρών μελών. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει έτσι ώστε χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Γαλλία που έχουν πολλά συμφέροντα στη νότια γειτονία να βοηθήσουν και αυτές οικονομικά, χρηματοδοτικά. Ε, να πω ότι εκπλήσωμαι ότι στην παρούσα φάση δεν ε, υποστηρίζουμε δράσεις στο κράτος του Ισραήλ. Όλοι γνωρίζουμε την κατάσταση η οποία δυστυχώς επικρατεί ε, ειδικά για την αραβική μειονότητα του Ισραήλ όπως επίσης και τους περιορισμούς τους οποίους θέτει ο νόμος για την λειτουργία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Λοιπόν, τι μπορείτε να κάνετε για τη χώρα αυτή, όπως επίσης και για την Αλγερία, χώρα στην οποία δεν θα επαρκώς. Ε, μία ερώτηση τώρα να μου επιτρέψετε να κάνω για τη Λευκορωσία. Ε, η Λευκορωσία δεν είναι προτεραιότητά μας ε, προς Ανατολάς τουλάχιστον. Ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι δεν σας επιτρέπουν ή δεν σας έχουν επιτρέψει τουλάχιστον μέχρι τώρα να ασχοληθείτε με την Λευκορωσία. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Μπουτικόφερ. Έχει έρθει είδα και ο συνάδελφος Μπροκ που είναι και αυτός μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος για τη Δημοκρατία. Βλέπω ότι οι ευρωβουλευτές έχουν μελετήσει πολύ καλά την ετήσια έκθεση που μας παρουσίασε ο Διευθυντής κύριος Πομιανόφσκι και τέθηκαν τα σημαντικότερα θέματα για την αποτίμηση αξιολόγηση του πρώτου χρόνου των εργασιών του. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να ζητήσω από τον κύριο Διευθυντή Πομιανόφσκι να μας κάνει μία σύντομη αλλά περιεκτική σύνοψη απάντηση των ερωτήσεων. Έχει 20 λεπτά. 20 λεπτά. 13 λεπτά με συγχωρείτε. Ευχαριστώ Πρόεδρε για τον γενναιόδωρο χρόνο που μου δίνετε 10 με 15 λεπτά. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα που τα βρήκα πολύ ενδιαφέροντα και θεμητά. Σας ευχαριστώ πολύ για όσα καλά λόγια είπατε για το Ίδρυμα. Είναι πολύ σημαντικό για όλους μας να έχουμε αυτή τη στήριξη εκ μέρους σας διότι είμαστε μικρή ομάδα και δουλεύουμε πάρα πολύ για να κατορθώσουμε ό,τι κατορθώσαμε. Πρώτα τα ερωτήματα. Τώρα τα ερωτήματα. Χριστιαν Πρέντα ρώτησε πώς θα εξισορροπήσουμε την ευληγησία με, με την αποτελεσματικότητα ώστε να χορηγούνται οργανωμένα οι δωρεές. Αυτά είναι τα μαθήματα που πήραμε και από την Ουκρανία γιατί πήγαμε στο Μαϊντάν και είδαμε σε επαναστατική, προεπαναστατική περίοδο και κοινωνική αναστάτωση ότι ακόμα και οι δικοί μας συντομότατη διαδικασία, ένα αίτημα τρισέλιδο αντί των εκατοντάδων σελίδων που χρειάζονται για τη χορήγηση ενωσιακών ταμείων. Ακόμη και αυτές οι τρεις σελίδες ήταν πολλές. Γιατί είναι και το θέμα της ε, νοοτροπίας του κόσμου ανάλογα με τη φάση στην οποία βρίσκονται κοινωνικά. Εκεί στο Μαϊντάν έλεγαν θέλουμε, θα ζητήσουμε τη στήριξή σας αλλά όχι από σήμερα. Όχι ακόμα γιατί δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε αύριο. Επομένως μπορεί να υπάρχουν καταστάσεις που ισχύουν μία μέρα και δεν μπορεί να μην ισχύουν την επόμενη. Όπως θα θυμάστε στο, στην Ουκρανία ο Γιαννουκόβιτς στις 16 Ιανουαρίου ε, θέλησε να εφαρμόσει ένα νόμο ανάλογο με τον του Πούτιν και της Αιγύπτου που απαγόρευε τις δραστηριότητες των μη κυβερνητικών οργανώσεων και μέσα σε μια νύχτα ή μέσα σε δύο μέρες <coughs> μπορούν να, μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα με τρόπο ο, πολύ σημαντικό μέσα σε μια νύχτα λοιπόν. Έτσι μάθαμε, αυτά τα μαθήματα πήραμε, ότι υπάρχουν καταστάσεις όπου πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει επαρκώς ευλίγιστη διαδικασία και υπάρχουν όρια για τα πάντα για την εξισορρόπηση μεταξύ πολύ εύκολων και ελαφρών διαδικασιών και της ευθύνης για την καλύτερη χρησιμοποίηση των ποσών. Και έρχομαι τώρα στο θέμα που έθεσε η κυρία Λόζινγκ πώς ξέρουμε σε ποιον να δώσουμε τα ποσά και τις δωρεές. Αυτό συνδέεται και με το ερώτημα του κυρίου Παντζέρη πώς διασφαλίζουμε την συνέργεια των διαφόρων προγραμμάτων που επιχορηγούμε. Βασιζόμαστε στην αρχή ότι πρέπει από την πρώτη μέρα να διασφαλίσουμε κοινέ πρακτικές. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε αποτελεσματικοί από τις Βρυξέλλες αν δεν έχουμε επαρκή συνεργασία με εκείνους που βρίσκονται επιτόπου εδώ και χρόνια. Εγώ φοβόμουν στην αρχή μήπως δεν υπάρξει αυτή η συνέργεια αλλά τελικά είναι από το πιο επιτυχές μέρος της, ε, του απολογισμού μας. Και οι πρεσβείες των χωρών μελών και οι αντιπροσωπείες της Ένωσης συνεργάστηκαν και τις πληροφορίες που μας χορηγούν τις συνδυάζουμε για να διασφαλίσουμε ότι αυτοί τους οποίους στηρίζουμε δεν θα είναι τυχαίοι. Και αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι μπορεί κάποιος να επιχορηγηθεί, κάποιος που δεν έκανε τίποτε ποτέ χθες και σήμερα βρίσκεται στο προσκήνιο. Γιατί εδώ χρησιμεύει ένα τέτοιο όργανο σαν το δικό μας. Όποιος, όποια μη κυβερνητική οργάνωση αποφασίσει από ουδετερότητα να περάσει στη δράση μπορεί να χρηματοδοτηθεί αν αποδείξει τη χρησιμότητα που έχει στην κοινότητά της. Μέχρι τώρα τα χέρια και τα βασικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ήταν έτοιμα για να υποστηρίξουν τη μετάβαση από επίπεδο ΜΚΟ σε επίπεδο πολιτικής δράσης. Τώρα το Ίδρυμα αυτό καλύπτει αυτό το κενό και δίνει υποστήριξη εκεί που δεν μπορούσε να δοθεί υποστήριξη στο παρελθόν. Χρειάζεται λοιπόν ταχύτητα, αλλά πρέπει να έχει κανείς μια σωστή επαφή για να συνεχίσει το έργο των τωρινών εργαλείων. ισορροπία μεταξύ Ανατολής και Νότου. Υποστηρίζω αυτά που είπε η κυρία Φωτίγκα για το θέμα αυτό. Δεν βλέπουμε κανένα τέτοιο πρόβλημα στο Ίδρυμα μας. Όπως βλέπετε στον πίνακα για τις ταπάνες μας ήταν 50-50 τα 100 η κατανομή Νότου και Ανατολής. Δεν βλέπουμε λοιπόν ως αντίμαχες τις δύο αυτές περιοχές, προσπαθούμε να τις καλύψουμε και τις δύο. Έχουμε μία, ε, μία ανάδραση επί τη βάση και των αιτήσεων που παίρνουμε. Η δημοκρατία δεν μπορεί να εξαχθεί, η δημοκρατία μπορεί να επιτευχθεί μονάχα με τον αγώνα αυτών που βρίσκονται στις τοπικές κοινωνίες. Και από αυτή την άποψη κατανοείται γιατί η Αλγερία έχει τόσο μικρή εκπροσώπηση στα προγράμματά μας. Γιατί παίρνουμε πολύ λίγες αιτήσει από την Αλγερία. Για μας λοιπόν είναι ένας πολύ δύσκολος εταίρος η Αλγερία. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανένα από την Αλγερία να ζητήσει υποστήριξη. Για το Ισραήλ και τη Ρωσία καταγράφω αυτό το οποίο ζητήσετε. Κατανοώ την επιχειρηματολογία σας. Το Διοικητικό μα Συμβούλιο έχει συζητήσει τα θέματα της διεύνησης τη γεωγραφική μας έντολη, αλλά αυτό βέβαια δεν εξαρτάται από τη γραμματεία, εξαρτάται από το Ταμείο, στο οποίο εκπροσωπήσετε κι εσείς. Μπορείτε λοιπόν να περάσετε αυτές τι ιδέες από τον μηχανισμό του ε, Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Για τη Λευκορωσία. Η Λευκορωσία φυσικά αποτελεί τμήμα των δραστηριοτήτων μας, αλλά στην Λευκορωσία έχουμε μια ιδιαίτερα δυσχερή κατάσταση εδώ και 20 χρόνια έχουμε τον ίδιο δικτάτορα και όλο αυτό το διάστημα έχουμε και την ίδια αντιπολίτευση. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να βρούμε νέους αναδυόμενους εταίρους. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τις υφιστάμενες ομάδες, αλλά ήδη έχουν μια επαρκή διεθνή υποστήριξη και είναι αναγνωρισμένοι στον τομέα αυτό. Επομένως, ο ρόλος του Ιδρύματος που οστιάζει στην ευέλικτη χρηματοδότηση δεν είναι τόσο κέριος για τη δραστηριότητα των ε, ομάδων της αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία. Γι' αυτό στη Λευκορωσία εμείς προσπαθούμε να δούμε νέους ηγέτες, νέες ομάδες ε, ακτιβισμού και ακόμα δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Η κατάσταση στην Ουκρανία βέβαια τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα για την κοινωνία της Λευκορωσίας βλέποντας τις δυσκολίες που ε, λαμβάνονται χώρα στην Ανατολική Ουκρανία και την ρωσική επιθετικότητα, βασικά φοβάται να μην αντιμετωπίσει μια αντίστοιχη κατάσταση και εμπόλεμες συνθήκες στη Λευκορωσία. Αυτά μας λένε οι ε, επιτόπια εργαζόμενοι ότι υπάρχει ακόμα λιγότερη προσπάθεια από την τοπική κοινωνία έναντι του παρελθόντος. Για τη διαφάνεια φυσικά εμείς θέλουμε να υπάρχει μια εξωτερική διαδικασία ελέγχου. Είχαμε μια ένα λογιστικό έλεγχο από την Κομισιόν, είχαμε και ένα θεσμικό έλεγχο που ζητήσαν ορισμένοι από τους χρηματοδότες μας και φυσικά τηρούμε όλους τους λογιστικούς κανόνες που εμπίπτουν στο βελγικό δίκαιο, διότι είμαστε ε, ένα ίδρυμα που υπόκειται στο, ελβε... στο βελγικό δίκαιο. Κάθε έξι μήνες επίσης δίνουμε μια λεπτομερή έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τις χρηματοδοτήσεις μας Γι' αυτό έχουμε και τόσο συχνές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι κάτι το χρονοβόρο για τη γραμματεία μας. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον δύο εβδομάδες για να προετοιμάσουμε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τουλάχιστον μία εβδομάδα χρειάζεται για να συντάξουμε τις απαραίτητες ε, εκθέσεις. Αυτό είναι απαραίτητο όμως για να έχουμε διαφάνεια και καλή δυνατότητα εποπτείας από το Διοικητικό Συμβούλιο. Και επίσης έχουμε φυσικά την Εκτελεστική Επιτροπή με έξι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ελέγχουν τις καθημερινές δραστηριότητές μας και φυσικά παρακολουθούν τα σχέδια εργασίας και τις δαπάνες μας. Από την άποψη αυτή τόσο ο θεσμικός έλεγχος όσο και η καθημερινή εποπτεία και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων μας έχει εξασφαλιστεί από τις διοικητικές μας δομές λιγότερο από 20% τώρα των σχεδίων μας έχουν το καθεστώς της χαμηλής ορατότητος. Και αυτό γίνεται στην περίπτωση που ένας δικαίουχος μπορεί να, είναι, να κινδυνεύει να φυλακιστεί ή να στιγματιστεί στην κοινωνία που βρίσκεται. Έχουμε λοιπόν δικαιούχους στη Συρία για προφανείς λόγους, όμως δεν θέλουμε να δώσουμε δημοσιότητα στην υποστήριξη που δίνουμε σε αυτούς. Το ίδιο συμβαίνει και στη Λευκορωσία και το ίδιο συμβαίνει στην Αίγυπτο. Το ερώτημα είναι πώς γίνεται κάτι τέτοιο και εδώ μπορώ να σας δώσω τη δική μου εμπειρία από τη δεκαετία του 1980 όταν ήμουν νεαρός ακτιβιστής στην πολωνική αντιπολίτευση χρησιμοποιούμε ακριβώς την ίδια τεχνολογία που είχαμε τότε. Θα το δείτε σε πολλά βιβλία και απομνημονεύματα. Πολλές φορές Απλώς με ένα φάκελο μπορούν να δίδονται αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Υπάρχει ο μηχανισμός λοιπόν εσωτερικού ελέγχου, αλλά βασίζεται και σε δεσμούς εμπιστοσύνης με ακτιβιστές που ρισκάρουν τη ζωή και την ελευθερία τους για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και πάντα γίνεται αυτό σε καταστάσεις όπου έχουμε τη διαβεβαίωση ότι πρόκειται για άτομα τα οποία είναι πραγματικοί αγωνιστές. Γίνονται αυτά λοιπόν επιλεκτικά και με καλή προετοιμασία. Εκεί όμως το, το πρωτεύον είναι η προστασία της ασφάλειας του δικαιούχου και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει και όλες οι διαδικασίες μας ευθυγραμμίζονται με αυτή την βασική πρώτη προτεραιότητα. Δεν ξέρω αν απάντησα όλα τα ερωτήματά σας, ίσως όχι, αλλά ο χρόνος δεν μου επιτρέπει να το πράξω. Σύμφωνα όμως με τον κύριο Παντσέρη, ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στις κέρδιες προτεραιότητές μας και φυσικά οι συνέργειες είναι απαραίτητες με όλα τα άλλα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία χρηματοδοτούν την κοινωνία των πολιτών και την ε, προστασία της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμείς όμως θέλουμε να καλύψουμε τα κενά τα οποία δημιουργούνται και να χρηματοδοτήσουμε εκεί πέρα που δεν μπορούν να δράσουν αυτά τα εργαλεία όταν έχουμε μη καταγεγραμμένες ομάδες, πολιτική δραστηριότητα και ταχεία αντίδραση που δεν μπορούν τα άλλα εργαλεία να την εξασφαλίσουν λόγω της διαδικασίας υποβολών προσφορών που μπορεί να, να καταδαπανίσουν πολύ χρόνο. Σταματώ λοιπόν εδώ. Με χαρά θα έρθω και πάλι ενώπιον σας αν απαραίτητο για να αντιμετωπίσω τα ερωτήματα που μπορεί να γεννηθούν στο μυαλό σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πομιονόσκη πολύ περιεκτική παρουσίασή σας. Ευχαριστώ όλους, όλα τα μέλη που συμμετέσχουν. Θα γίνει ένα μονόλεπτο διάλειμμα τώρα και θα συνεχίσει να προεδρεύει ο πρόεδρος Μπροκ για την επίσκεψη του κυρίου Μπαρζάνη επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιρακινού Κουρινιστάν. Meine Damen Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, συγγνώμη που καθυστέρησα να έρθω στη συνεδρίαση, αλλά έχει μόλις λάβει η χώρα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Κινέζων Κομμουνιστών στην οποία έπρεπε να συμμετάσχω. Έχουμε τώρα όμως την ε, συνάντηση με τον κύριο ε, Μπαρτσάνη, τον επικεφαλή Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιρακικού Κουρδιστάν. Καλώς ήρθατε κύριε Μπαρτσάνη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και για την παρουσία σας και μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτά τα οποία θα μας πείτε. Χαιρόμαστε για την παρουσία σας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και μας ενδιαφέρει πολύ η άποψη της κυβέρνησης του Ιρακινού Κουρδιστάν ε, σε σχέση με τον αγώνα κατά του Ισλαμικού Χαλιφάτου. Γνωρίζουμε τα γεγονότα στο Κομπάνι, η διεθνής κοινότητα έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να έρθει μια πρώτη ομάδα από Ιρακινούς μαχητές για την ανακούφιση του κομπάνι και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε περαιτέρω πόρους για κάτι τέτοιο. Θα διασχίσουν την Τουρκία για να φτάσουν στο κομπάνι οι <clears throat> αγωνιστές αυτό είναι σημαντικό για να έχουμε ένα δρόμο ενίσχυσης του κομπάνι στο μέλλον. Ξέρω ότι οι συμπολίτες σας έχουν αναλάβει σημαντικές ευθύνες για την υποστήριξη των Κούρδων ε, φίλων σας στο Κομπάνι. Θέλω να σας ευχαριστήσω όμως επίσης και για αυτά που κάνατε για να προστατεύσετε τους Γέζιντι και άλλους στην δική σας περιοχή του Ιράκ και τις μεγάλες ευθύνες που έχετε αναλάβει. Ξέρουμε όλοι πόσο είναι δύσκολη η κατάσταση. Γίνεται ένα είδος πολέμου δια αντιπροσώπων και υπάρχει ένα εκρηκτικό μείγμα σε πολιτικό και θρησκευτικό επίπεδο και εμείς δεν γνωρίζουμε πάντα την πραγματικότητα εδώ στην Ευρώπη. Ίσως μπορείτε να μας βοηθήσετε να έχουμε μια καλύτερη πληροφόρηση η οποία θα μας επιτρέψει να φέρουμε σε πέρας και το δικό μας ε, εγχείρημα του να αποτρέψουμε τις γενοκτονίες σε αυτό το τμήμα του κόσμου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε Ελμπερμπρόκ, Κύριοι βουλευτές της Επιτροπής Εξωτερικών κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να παρουσιάσω την κατάσταση από απόψε ασφαλείας στο Ιρακινό Κουρδεστάν. Βρισκόμαστε εδώ σε εποχή κρίσιμη για τους λαού της Μέσης Ανατολής και γενικότερα της διεθνούς κοινότητας. Σημειώνονται όλο και περισσότερα αθώα θύματα που σφαγιάζονται, αποκεφαλίζονται στο Ιράκ και τη Συρία και αυτό σοκάρει τις συνειδήσεις του ελευθέρου κόσμου. Πολλές χώρες έχουν θελήσει να λάβουν ύψης του επίπεδου μέτρα ασφαλείας. Είναι λοιπόν μια περίοδος πολύ προκλητική και δύσκολη για την διασφάλιση διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Η διεθνής κοινότητα όμως φαίνεται να μην είναι και τόσο πρόθυμη να πάρει τις αποφάσεις που αρμόζουν για να προστατευτούν οι ζωές τόσων αυτών. Αυτή, αυτή η διστακτικότητα επέτρεψε την, ε, στο ίσις να μπει στο κομμάτι στο Ιράκ και στη Συρία και να σφάξει τόσους ανθρώπους σε επίπεδα γενοκτονίας. Σήμερα το Ιρακινό Κουρδιστάν δεν πολεμούμε μόνο για την ανεξαρτησία μας όπως καθόλου τον 20ο αιώνα αλλά υπέρ όλου του ελεύθερου κόσμου. Στις 8 Ιουνίου, δύο μόλις μέρες πριν πέσει η Μοσούλη στο χέρια του Ίσης, πληροφορήσαμε την Ιρακινή κυβέρνηση ότι πρόκειται να γίνει επίθεση και προσφέρθηκαν οι Πεσμεργά να προστατεύσουν την πόλη. Αντί, α, δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Και δύο μέρες αργότερα μπήκαν στη Μοσούλη οι μαχητές του Ίσης και κατέλαβαν τις κέρυες στρατηγικές θέσεις της πόλης και τα κυβερνητικά κτίρια. Ταυτόχρονα κατέρεε η επίσημη στρατιωτική Ιρακινή άμυνα και τις επόμενες ώρες πέντε μεραρχίες Ιρακινές τελείως υποχώρησαν και διαλύθηκαν και μπόρεσαν οι μαχητές του Ίσης να πάρουν τα βαρέα όπλα τους και τα ελαφρά. Και έτσι καταλήξαμε στη δημιουργία ενός τρομοκρατικού ψευτοκράτους το οποίο στο εξής διαθέτει και τάγκς και όλμους και βαριά όπλα. Όπλα τα οποία έχει αρπάξει από το στρατό στο Ιράκ αλλά και από τη Συρία. Το ίσις χρησιμοποίησε πολλά τέτοια όπλα και μαχητές για να τρομοκρατήσει ολόκληρα χωριά, μειονότητες και οικογένειες. Δεκάδων χιλιάδων χριστιανών και γεζίδι αναγκάστηκαν να στραφούν στο Ισλάμ με το ζόρι. Και χιλιάδες οικογενειών άρχισαν να αντιμετωπίζουν μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Στις 3 Αυγούστου το Ίσις κατέλαβε και την πόλη της Χορτάν. Είμαστε ευγνώμονες προς τις Ηνωμένε Πολιτείες και τις ευρωπαϊκές χώρες γιατί άκουσαν επιτέλους τις εκκλήσεις μας για αεροπορική υποστήριξη αλλά χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες. Στο Σιντζάρ έγιναν τρομερές βιοπραγίες. Γείτονε που ζούσαν ειρηνικά επί πολλές γενιές στράφηκαν κατά τον Γεζίντιε. Σημειώθηκαν πάρα πολλές δολοφονίες και δεκάδες χιλιάδων Κούρδων αναγκάστηκαν να φύγουν στα βουνά. Κάτω από τον καυτό ήλιο χωρίς τρόφιμα και νερό συνέχισαν να φεύγουν ενώ τους κυνηγούσαν οι μαχητές του Ίσις. Α, εδώ πρόκειται για γενοκτονία κατά των Κούρδων και των Γεζίδη. Και είναι κάτι που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί και προβλεφθεί. Οι ρήψει υλικού στα βουνά από αεροπλάνα έσωσαν πολλές ζωές. Αλλά βέβαια υπάρχουν ακόμη πολλοί που πολλούνται ως δούλοι σε αραβικές φυλές και εμείς έχουμε υποστεί εθνοκάθαρση και γενοκτονία καθώς και υποστεί τη χρήση χημικών όπλων. Έχουμε καταφέρει να πάρουμε πίσω ορισμένα κομμάτια της γης που μας έκλεψε το ίσις αλλά δεν τελειώσε ο αγώνας. Οι στρατιωτικές ικανότητες, δυνατότητες του ίσις θα είναι ο φασιστικός παράγοντας γιατί έχουν πολλή χρηματοδότηση από χώρες της Μέσης Ανατολής και αλλού. Δεν αναγνωρίζουν σύνορα και δεν θα διστάσουν να επιτεθούν όποτε και όπου μπορούν. Για να το θέσω έτσι γενικότερα, το ίσις διαθέτει 3 με 6 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο με την ε, λαθροπόληση πετρελαίου στη μαύρη αγορά. Επίσης παίρνει τρόφιμα δημητριακά και φορολογεί τον κόσμο που έχει κατακτήσει. Έχει προωθημένα όπλα και διαθέτει χιλιάδες ξένων μαχητών και από ευρωπαϊκές χώρες που σπέβδουν στη Μέση Ανατολή για να πολεμήσουν με το ίσις. Και αυτό δεν απειλεί μόνο το Κουρδιστάν αλλά όλες τις χώρες της περιοχής και τις δυτικές χώρες. Ήδη έχουμε δει ότι γίνονται διαδηλώσεις υπέρ του σε, και σε ευρωπαϊκές πόλεις. Μην νομίζετε λοιπόν ότι είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον αγώνα. Πρόκειται για κοινό εχθρό και κοινή ευθύνη. Το Κουρδιστάν δεν καταπολεμά μόνο τους τζιχαδιστές αλλά τρομοκράτες και από ευρωπαϊκές χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο και πολλές άλλες που έχουν αποφασίσει να μας σκοτώσουν όλους. Δεν μπορούμε να έχουμε, διαπραγματευτούμε μαζί τους, δεν καταλαβαίνουν τι θα πει συνύπαρξη, ειρήνη, δημοκρατία, δεν, δεν έχουμε κοινέ αξίες. Η ηρωική Πεσμεργά είναι στην πρώτη γραμμή αυτή τη στιγμή για την καταπολέμηση των τρομοκρατικών οργανώσεων που είναι αποφασισμένες να φέρουν το χάος και την καταστροφή στη Μέση Ανατολή. Οι πεσμεργά μας καταπολεμούν έναν εχθρό που διαθέτει πλήρη υλικό κράτους, ενός πλήρους κράτους, ολόκληρου κράτους. Εμείς λοιπόν πολεμάμε υπέρ του ελεύθερου κόσμου, αλλά ο ελεύθερος κόσμος με τη σειρά του δεν θέλει να μας βοηθήσει και να μας διαθέσει τα μέσα που χρειαζόμαστε για να προστατεύσουμε και τον κόσμο αυτόν και το λαό μας. Στις 25 Οκτωβρίου τρία, τρεις γενναίοι αδελφοί σκοτώθηκαν μαρτυρικά από το Ίσης. Μπορεί να μην γνωρίζετε τα ονόματά τους αλλά εμείς δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ γιατί σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα μιας ε, επίθεσης αυτοκτονίας διότι δεν είχαν τα όπλα που χρειάζονταν που να μπορούν να διαπεράσουν λαμαρίνες αυτοκινήτων. Και όλα αυτά γίνονται ενώ ο υπόλοιπος κόσμος παρατηρεί χωρίς να αντιδράει. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να ενισχυθεί ο αγώνας εναντίον του Ισλαμικού κράτους και γι' αυτό είμαι ενώπιον σας. Σήμερα το Ιρακινό Κουρδιστάν αγωνίζεται εναντίον τριών αντιπάλων. Καταρχήν είναι ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας. Είναι η ISIS τώρα, αλλά ήταν η Αλκάιντα στο παρελθόν. Το καθεστώς Μπαθ και άλλες κυβερνήσεις έχουν χρησιμοποιήσει χημικά όπλα εναντίον του λαού μας και έχουν καταστρέψει πάνω από 4.500 χωριά. Έχουμε αγωνιστεί εναντίον της τρομοκρατίας, εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε και να προασπίσουμε το λαό μας. Δεύτερον, έχουμε να κάνουμε ένα οικονομικό πόλεμο με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στη, του Ιράκ. Ένας από τους λόγους που δεν είχαμε αρκετά όπλα εναντίον του ISIS ήταν γιατί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν δίνει εξοπλισμό ούτε εκπαίδευση ούτε όπλα στους Πεσμεργά παρά τις συνταγματικές της υποχρεώσεις. Οι Πεσμεργά γνωρίζουν ότι είναι καθήκον τους να αγωνιστούν και να πεθάνουν για το Ιράκ αλλά τα δικαιώματά τους δεν λαμβάνονται υπόψη. Παράνομα η κυβέρνηση του Ιράκ έχει αναστείλει την μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων και του στρατού μας από το Φεβρουάριο του 2014 και οι Πεσμεργά εξακολουθούν να αγωνίζονται κατά τη τρομοκρατίας χωρίς υποστήριξη από την Ιρακινή κυβέρνηση και χωρί μισθοδοσία. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά έχουμε περιορισμένους πόρους. Είμαστε οι μόνοι οι οποίοι έχουμε κερδίσει έδαφο εναντίον τη ISIS, αλλά δεν έχουμε βαρέα όπλα από την Βαγδάτη ούτε από τους ε, συμμάχους μας στον διεθνή συνασπισμό εναντίον του ISIS. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο εκτοπισμένους και πρόσφυγες στο έδαφος μας και αυτό περιορίζει τη δυνατότητά μας να τους φροντίσουμε. Εμείς δίνουμε τη φιλοξενία μας στα άτομα αυτά χωρίς κανένα οικονομικό αντιστάθμισμα από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση του Ιράκ. Και τρίτον και πιο σημαντικό, η κυβέρνηση του Ιράκ εξακολουθεί να πιέζει τις χώρες της Δύσης που μας δίνουν βοήθεια ανθρωπιστική και όπλα, ζητά όλες αυτές οι αποστολές να περνούν από τη Βαγδάτη και αυτό καθυστερεί την παραδοσή τους. Με τον τρόπο αυτό χάνονται ζωές στο μέτωπο και τίθενται σε κίνδυνο οι ζωές αυτών που πρέπει να υποστηριχθούν. Και έρχομαι τώρα στο τελευταίο πιο σημαντικό στοιχείο. Κάνουμε ένα πόλεμο για μεγαλύτερη υποστήριξη από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δύσης. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε τον πόλεμο με Καλάσνικοφ και ε, εκτοξευτές χειροβομβίδων. Πρέπει να έχουμε βαρύτερα όπλα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις, ε, ε, τα βαρέα όπλα και τα άρματα μάχης. Μας είπαν ότι δεν μπορούμε να έχουμε λόγω της Βαγδάτης υποστήριξη σε βαρέα όπλα για τους Πεσμεργά. Αυτή είναι μια λαθασμένη πολιτική και πρέπει να αναθεωρηθεί. Υπήρξαν κάποιες γενναιόδορες χορηγίες από ευρωπαϊκές χώρες, αλλά ήταν κυρίως ελαφρά όπλα και πυρομαχικά. Δεν μπορούμε όμως να αντιμετωπίσουμε ένα οργανισμό που έχει τεράστια ε, εισοδήματα από το λαθρέμπορο, από το λαθρεμπόριο πετρελαίου και να τους αντιμετωπίσουμε μόνο με ελαφρά όπλα. Βάσει του συντάγματος του Ιράκ η ασφάλεια της ε, περιοχής του Ιρακινού Κουρδιστά εναπόκειται στους Πεσμαργά. Εμείς έχουμε αποφασίσει το 2003, είχαμε αποφασίσει να είμαστε τμήμα ενός νέου ανεξάρτητου Ιράκ μετά από την ε, κατάρρευση του καθεστώτος του Σαντάμ Χουσέιν. Και έχουμε αγωνιστεί για το να καταστραφεί αυτό το καθεστώς. Στείλαμε δυνάμεις στη Βαγδάτη το 2003 και 2006 για να καταστήλουμε τις ταραχές κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου που λάμβανε χώρα τότε. Αλλά πρέπει και το Ιράκ να αναλάβει τι ευθύνε. του. Είναι απαράδεκτο η Βαγδάτη να περιορίζει τη χρηματοδότηση του τμήματος του Ιρακινού Κορδιστάν λόγω της ε, διαφωνίας που έχει με μας και να μην δίδει βαρύ εξοπλισμό στους Πεσμεργά. Μπορεί η ISIS να νικηθεί μονάχα αν όλοι αναλάβουν τις ευθύνες τους και αυτό περιλαμβάνει το Ιράκ και τις γειτονικέ χώρε. Είμαστε έτοιμοι να, να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και τις διαφορές μας με τη Βαγδάτη με ειδικό τρόπο, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί το σημερινό status quo. Έχουμε τονίσει και έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν ότι είμαστε ένα λογικό και επικοδομητικό στοιχείο υπέρ της ασφάλειας και της ειρήνης στο διεθνή χώρο. Το να σταματήσει το χάος και η βία στο Ιράκ θα πρέπει να επιτευχθεί με την υποστήριξη του Κουρδιστάν. Η σταθερότητα στο Ιράκ έχει σημασία και για τη δική μας ασφάλεια. Η διεθνής τρομοκρατία πρέπει να αντιμετωπιστεί με διεθνή απάντηση και το Κουρδιστάν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Τώρα πια πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει ένα ηγετικό ρόλο και να αναβαθμίσει την υποστήριξη προς εμάς. Ο στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τη δημοκρατία στο Ιρακινό Κουρδιστάν και να διατηρήσουμε τις τοπικές του κοινότητες. Αλλά πρέπει η διεθνής κοινότητα να δώσει υποστήριξη στους γενναίους Πεσπερμά πεσμεργά. Το Ιρακινό Κουρδιστάν χαίρεται που μπορεί να υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την ειρήνη και την ελευθερία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως θα πρέπει να συνεργαστεί μαζί μας για να μπορέσει να κατατήσει μια στρατηγική με την οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί και να νικηθεί η τρομοκρατική απειλή για να μην έχετε να την αντιμετωπίσετε εδώ στις πρωτεύουσές σας. Δεν υπερασπίζουμε μονάχα τον κουρδικό λαό, αλλά και εκατομμύρια που ανήκουν σε άλλες εθνοτικές και ε, θρησκευτικές πρέπει να βοηθήσουμε όλους αυτούς οι οποίοι είναι θύματα καταδίωξης και καταστολής στο Ιράκ και αλλού. Έχουμε αναπτύξει πεσμέργα στο κομπάνι για να βοηθήσουν τους ομοφίλους του της Συρίας που αγωνίζονται για την προστασία αυτής της πόλης. Η κυβέρνησή μας και οι θεσμοί μας περιλαμβάνουν ανθρώπους από όλες τις κοινωνικές και εθνοτικές ομάδες. Είναι μια εμπειρία η οποία έχει λειτουργήσει για πάρα πολλούς αιώνες στην κουρδική ιστορία. Είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε. Η εμπειρία μας βασίζεται στην αρχή του σεβασμού για την ανθρώπινη ζωή και τη συνύπαρξη. Δεν είμαστε απειλή για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Είμαστε ακριβώς μια όαση ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή αυτή μέσα στο χάος και την αβεβαιότητα. Εν κατακλείδη και εξ ονόματος του, της κουρδικής περιοχής του Ιράκ θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της για τη συνεχή ανθρωπιστική βοήθεια που δίνει στα, στις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων που ζητούν καταφύγιο στην περιοχή μας. Βλέπουμε αισιόδοξα το μέλλον και προσβλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περαιτέρω υποστήριξή της. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και πάλι που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να λάβω το λόγο ενώπιόν σας και είμαι έτοιμος να απαντήσω στα ερώτηματά σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πεγιόν έχει πρώτος το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Μπαρζανή για την ειλικρίνεια που χαρακτήρισε την παρέμβασή σας. Μιλήσατε με λόγια σκληρά απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την διεθνή κοινότητα. Όπως επίσης μιλήσατε και με ακόμα πιο σκληρά λόγια για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Ιράκ που δεν σας στηρίζει στον δίκαιό σας αγώνα. Τρεις ερωτήσεις οι οποίες συνδέονται με το γενικότερο περιβάλλον. Από τη μία διακρίνουμε ξεκάθαρα ότι ο πόλεμος εναντίον του ε, Ισλαμικού κράτους δημιουργεί στρατηγικές αλλαγές στην περιοχή. Αυτό τροποποιεί τη σχέση σας με την Τουρκία η οποία ήταν διστακτική ε, στη βοήθεια προς τους Κούρδους μαχητές. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο βλέπετε τον συσχετισμό δυνάμεων ε, γύρω σας. Ο Μασούτ Μπαρζανί, ο πρόεδρος, ζήτησε να υπάρξει ένα δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία του Ιρακινού Κουρδιστάν. Τι γίνεται με το δημοψήφισμα αυτό. Πώς βλέπετε ε, την κατάσταση επίσης στο Κυρκούκ και κλείσατε με το τελευταίο θέμα. Σήμερα βλέπουμε πεσμεργά οι οποίοι προέρχονται από το κόμμα 5 και άλλοι από το κόμμα 5K. Πώς ακριβώς συνεργάζεστε μεταξύ σας και ε, πώς μπορούμε να είμαστε κι εμείς αισιόδοξοι όπως είπατε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κυρία Λιώ Μαρή, σας ευχαριστώ για την εξαιρετική και πληρέστατη παρουσίασή σας. Ε, κάποιες ερωτήσεις σχετικές με την ισορροπία δυνάμεων. Καταρχάς για τους Πεσμεργά, ε, αριθμητικά πόσοι είσαστε σε σχέση με τις δυνάμεις του Ισλαμικού κράτους. Ένα από τα, πλεονεκτήματα τα οποία έχετε είναι η γνώση της περιοχής και του αναγλήφου της ε, Έχετε κάποιο σύστημα ενημέρωσης ε, για το τι συμβαίνει στα εδάφη τα οποία έχει κατακτήσει το Ισλαμικό κράτος. Ε, και όταν ζητάτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να σας στηρίξει με συγκεκριμένα μέσα εσάς και τους μαχητές σας θα ήθελα να μάθω ποιοι είναι τελικά κατά σας οι τομείς του οποίους θεωρείτε ότι υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Μιλήσατε για βαρέα όπλα. μόνον αυτό. Αεροπορικά μέσα τι γίνεται. Και οι μαχητές τους οποίους αναφερθήκατε έχουν την καρτάρτιση που απαιτείται έτσι ώστε να χειριστούν αυτά τα μέσα τα οποία έχετε ανάγκη. Ο κύριος Τάνοκ. Κύριε Μπαρσάνη, καλώς ήλθατε και εγώ θέλω να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία να σας χαιρετήσω εξ ονόματος της ομάδας των συντονιστών ως συντονιστής της ομάδας αυτής και να χαιρετήσω και το θάρρος των ε, Πεσμεργά εναντίον του Ισλαμικού κράτους σε ένα αγώνα επιβίωσης για την δική σας περιοχή αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την τεράστια μάστιγα. Πιστεύω επίσης ότι η το Ισλαμικό Κράτο μπορεί να έχει κάνει εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητας και εγκλήματα γενοκτονία ενδεχομένω εναντίον το ESD και θα ζητήσω από τα Ηνωμένα Έθνη και όλα τα αρμόδια όργανα να εξετάσουν αυτό το στοιχείο. Χαίρομαι για το γεγονό ότι έστω και εκ των υστέρων η Τουρκία δέχτηκε να δώσει ελεύθερη διέλευση στους Πεσμεργά προ το Κομπάνι και ξέρω τώρα ότι αγωνίζονται μετά μαζί με τους τοπικούς μαχητές για να προασπίσουν την περιοχή αυτή. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σας για τις συνευτικές συνομιλίες μεταξύ της Άγκυρας και του κ. Ετζαλάν και την αναθέρμανση της διαδικασίας ειρήνευσης ε, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν προβλήματα με την διέλευση των αγωνιστών προς το κομπάνι το τελευταίο καιρό. Θεωρείτε ότι είναι καιρό να αναθεωρηθεί ο χαρακτηρισμό του ΠΚΚ ω τρομοκρατική οργάνωση. Επίση, θεωρείτε ότι οι χώρε του Περσικού κόλπου όπω το Κατάρ έχουν σταματήσει κάθε χρηματοδότηση προ του τζιχαδιστέ, γιατί ένα τμήμα αυτή τη χρηματοδότηση μπορεί να έχει φτάσει στα, στην ISIS. Πιστεύω ότι η περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν έχει σταθεί φάρο σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή και χρειάζεται όλη την υποστήριξή μα και ελπίζω ότι η νέα κυβέρνηση του Αλαμπάντ στην ε, Βαγδάτη που έχει ένα Υπουργό Οικονομικών από την Κουρδική Συνιστόσα θα μπορέσει να συνενώσει όλες τις κοινότητες του Ιράκ και να διαμοιράσει ισοδίκαια τους πόρους που πρέπει να έχει και η δική σας περιοχή που μέχρι τώρα σας τις είχαν αρνηθεί. Σας ελπίζω λοιπόν, σας εύχομαι μάλλον μια επιτυχή επίσκεψη Βρυξέλλες και στα ευρωπαϊκά όργανα. Κυρία Σάκη, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Μπαρζάνη για το γεγονό ότι είναι μπροστά μα και συζητά μαζί μα σε αυτέ τι δύσκολε συνθήκε και για εσά αλλά και για το όλο κόσμο. Φοβάμαι ότι η Μέση Ανατολή έχει υποφέρει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από την έννοια, από την ιδέα ότι ο εχθρό του εχθρού μου είναι φίλος μου. Θα ήθελα να σας ζητήσω να μας πείτε πώς βλέπετε το ρόλο του Ισλαμικού κράτους του Ιράν σε ό,τι αφορά τον αγώνα κατά του Ισλαμικού κράτους της Συρίας και της Ανατολής και επίσης την επιρροή που μπορεί να έχει πάνω στη Βαγδάτη και αν μπορείτε να μας πείτε επίσης κάτι περισσότερο σε σχέση με τις συνομιλίες μεταξύ Τουρκίας και Κούρδων. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Λέζιν, κύριε Μπατσάνη. με στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το γεγονός ότι η αντίσταση κατά των ομοτήτων του φασιστικού Ισλαμικού κράτους θα πρέπει να ενισχυθεί. Και πάλι θέλω να στέσω αυτό το ερώτημα. Πώς βλέπετε το ρόλο του ΠΚΚ στον αγώνα αυτό. Πώς αντιμετωπίζετε την αίτηση αυτή να ανοίξει η Τουρκία τα σύνορά της στους μαχητές του ΠΚΚ Επίσης έχετε παίξει ένα σημαντικό ρόλο για τη διάσωση των Γεζιντή και την ε, προστασία της Βόρειας Συρίας, της Ροζαβά. Ποιες είναι οι απόψεις σας για την παράδοση δυτικών όπλων στους μαχητές της ε, Ροζαβά του Συριακού Κουρδιστάν Ποιες είναι οι θέσεις λοιπόν για το αν πρέπει να εξοπλιστούν αυτές οι ομάδες και πώς αντιμετωπίζετε και πάλι την, έννοια, την ιδέα αυτή ότι η Τουρκία θα ήθελε να δημιουργήσει ένα, μια ουδετεροποιημένη περιοχή στην βόρεια Συρία, στη Ρόζαβα. Επίσης, σε σχέση με την αποστολή Πεσμεργά στο, στη Βόρεια Συρία και το Κομπάνι. Θα ήθελα να ξέρω αν συνδέθηκε αυτή η αποστολή αγωνιστών σε κάποιες ε, ε, σε κάποια αντισταθμίσματα, σε κάποιες ε, απαιτήσει και πώς σε αυτή την συνολική αυτή κατάσταση και στον αγώνα εναντίον του Ισλαμικού κράτους βλέπετε το ρόλο του Μπασάρα Λασάντ. Είναι ο Μπασάρα Λασάντ ένας σύμμαχος σε αυτόν τον αγώνα ή εξακολουθεί να υποστηρίζει το Ιρακινό Κούρδισταν την υποστήριξη των ε, θέσεων που θέλουν μια αλλαγή κυβέρνησης στη Συρία. Ευχαριστώ. Thank you, President. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Μπαρζάνη, και εγώ θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή μας, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Είμαι πίσω από την τηλεοπτική κάμερα, δεν με βλέπετε. στηρίζω τα σχόλια των συναδέλφων που μίλησαν νωρίτερα. Αναφερθήκατε πιο συγκεκριμένα στο ότι το Ισλαμικό κράτος έχει ε, βγάλει από, τα, από τις πωλήσει πετρελαίου εκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα. Τι μπορούμε να κάνουμε όπως ακριβώς εμείς ασχολούμεθα με αντίστοιχες καταστάσεις στα λεγόμενα ματωμένα διαμάντια ή που έρχονται δηλαδή από περιοχές στις οποίες υπάρχουν πολεμικές σειράξεις. Τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να μειώσουμε τις δυνατότητες που έχουν α, ε, τις ε, δυνατότητες αγοράς όπλων ε, εμποδίζοντας τη λειτουργία των λεγόμενων κινητών δηληστηρίων τα οποία χρησιμοποιούν και θα ήθελα να δω τι γίνεται και με το καθεστώς του ΠΚΚ στην Τουρκία. Αυτό θα ήταν κάτι το χρήσιμο να συζητήσουμε. Ποια είναι η άποψή σας. Και επίσης να μας, δώσουμε, να μας δώσετε κάποιες περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό της κεντρικής κυβέρνησης της Βαγδάτης που έχει παγώσει τις πληρωμές και δεν αναφέρομαι στα όπλα αλλά σε επίπεδο λειτουργικής χρηματοδότησης. Είναι κάτι το οποίο ίσως μπορούμε να βοηθήσουμε με υψηλότερη από ό,τι τώρα ταχύτητα. Mr. Bazani, the Έχετε το λόγο κύριε Μπαζάνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Προσπαθήσω να απαντήσω όλα αυτά τα ερωτήματα που μου τέθηκαν με τον πιο συγκεκριμένο δυνατό τρόπο. Αν υπάρχουν ε, αλλαγές στις ε, ανάγκες μας, νομίζω το πρώτο ερώτημα το οποίο ετέθη είναι η σχέση μας με την Τουρκία και το τι περιμένουμε από την Τουρκία σε σχέση με τις ανάγκες που έχουμε και την υποστήριξη που χρειαζόμαστε σε ό,τι αφορά βαρύ εξοπλισμό. Πράγματι χρειαζόμαστε βαρύ εξοπλισμό. Χρειαζόμαστε εξελιγμένα όπλα για να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό μας. Είναι ένας εχθρός ο οποίος έχει καταλάβει, έχει πάρει όπλα από τον διαλυμένο Ιρακινό στρατό όταν αντιμετωπίσαν τους Πεσμεγά ήταν πολύ πιο καλά εξοπλισμένοι έναντι της εποχής που πολεμούσαν μονάχα τον Ιρακινό στρατό, γιατί ήρθαν μαζί με τον εξοπλισμό που κατέλαβαν από τον Ιρακινό στρατό. Είχαν πυράβλους, είχαν πυροβολικό μεγάλης εμβέλειας, είχαν αμερικάνικα χάμβις, είχαν πυρομαχικά, είχαν εξοπλισμό λοιπόν, ο οποίος ήταν πολύ ισχυρότερος από αυτόν που είχαν οι δικοί μας μαχητές οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να λειτουργούν με πεπαλαιωμένα ε, πολεμικά όπλα τα οποία είχαν αποκομίσει από τον προηγούμενο πόλεμο στο Ιράκ. Και αντί να έχει υποστήριξη από, τους, ε, από την κεντρική κυβέρνηση ο στρατός μας, όχι μόνο δεν είχε κάτι τέτοια υποστήριξη, αλλά δεν τους επέτρεψε να αποκτήσουν πιο σύγχρονα όπλα. Όταν μιλάτε λοιπόν για βαρύ εξοπλισμό, μιλάμε για βαρύ πυροβολικό, για άρματα μάχης, για θωρακισμένα οχήματα για να μπορούν οι Πεσμεργά να αντιμετωπίσουν εποφελώς την, ε, το Ισλαμικό κράτος, ελικόπτερα για να μπορέσουν να μεταφέρουν τους τραυματίες στα νοσοκομεία. Είναι όλα αυτά λοιπόν ο εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για να νικηθεί αυτός ο στρατός για την Τουρκία. Εμείς περιμένουμε ότι η Τουρκία θα είχε παίξει ένα πιο σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των Πεσμέργα και των συμμάχων εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Μας είπαν στην αρχή ότι γινόντουσαν οι προεδρικές εκλογές τότε στην Τουρκία και είχαν και το πρόβλημα των ομήρων της Μοσούλης που είχε στα χέρια της το Ισλαμικό κράτος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι στην αρχή θα μπορούσαν να είναι διστακτικοί για την συμμετοχή τους. Πάντα όμως ελπίζαμε και εξακολουθούμε να ελπίζουμε ότι η τουρκική βοήθεια θα είναι πολύ περισσότερη από αυτή που είχε σταθεί μέχρι τώρα για το δημοψήφισμα και το τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι δικαίωμα των Κούρδων να κάνουν ένα δημοψήφισμα <clears throat> για το μέλλον ορισμένων περιοχών. Πρέπει να ξέρουμε τι θέλει ο κουρδικός λαός για το μέλλον του. Η πρόταση δημοψηφίσματος πήγε στο κοινοβούλιο μας, το κοινοβούλιο μας την έχει αποδεχτεί και τώρα προετοιμάσουμε το δημοψήφισμα αυτό. Το να έχουμε ένα δημοψήφισμα είναι ένα πράγμα, το πώς θα εφαρμοστούν τα αποτέλεσματα του δημοψηφίσματος είναι κάτι διαφορετικό. Θέλουμε το δημοψήφισμα αυτό να γίνει με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε όλοι θα ξέρουν τι ακριβώς ζητά σε επίπεδο αυτοδιάθεσης ο λαός του Κουρδιστάν και πώς θέλει να αντιμετωπίσει το μέλλον του. Υπήρξε ένα ερώτημα για το αν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των ε, Πεσμέργα και των, δυνάμεων της, ε, των κουρδικών δυνάμεων της Βόρειας Συρίας. Όλα αυτά βρίσκονται στα μάλλον και των αγωνιστών των διαφόρων κομμάτων στο Κουρδιστάν. Το Υπουργείο Άμυνας είναι αυτό το οποίο συντονίζει όλες τις ενέργειες των Πεσμεργά και ελέγχει όλες αυτές τις ένοπλες δυνάμεις ανεξάρτητα από την πολιτική συνιστόσα και προέλευση που έχουν. Θέλουμε λοιπόν να ενσωματώσουμε όλες μας στρατιωτικές δυνάμεις. Αυτή είναι μια συνεχής ε, διαδικασία. Δυστυχώς το κάνουμε αυτό ενώ συγχρόνως πρέπει να αντιμετωπίσουμε το Ισλαμικό κράτος. Είναι μια μακρά μεταβατική λοιπόν διαδικασία που πρέπει να γίνει, αλλά σίγουρα θα ολοκληρωθεί εν καιρό. Πόσοι υπεσμέρκα υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Οι μάχημες δυνάμεις μας δεν είναι πολύ αυτοί οι οποίοι έχουν φέρει όπλα είναι περίπου 150.000 στην περιοχή του Κουρδιστάν. Δεν είναι όλοι τους μάχημες δυνάμεις και δεν είναι όλοι αυτοί αρκετά νέοι για να πάνε στην πρώτη γραμμή. Αυτοί οι οποίοι όμως πολεμούν είναι περίπου 40 με 60.000 εξαρτάται από πόσοι χρειάζονται σε κάθε μέτωπο και πώς μπορούν να αντικατασταθούν. Ο συνολικό αριθμό, όπω σα είπα, είναι περίπου 150.000 σε όλε οι ενόπλε δυνάμει μα Και πόσου αντιμετωπίζουν από, την, από το Ισλαμικό κράτο, από την ISIS. Η ISIS έχει τους ε, πιο σκληροτράχυλου μαχητέ, οι οποίοι είναι ίσω λίγοι, αλλά αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν την ISIS και έχουν ε, στρατολογηθεί από την ISIS στο Ιράκ και τη Συρία, ξεπερνούν τι 40.000. Είναι τουλάχιστον 18.000 στο Ιράκ και περίπου 22.000 στη Συρία πέραν αυτών υπάρχουν και οι διάφορες ε, φυλές, τοπικές φυλές που υποστηρίζουν την ISIS. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί οι οποίοι υποστηρίζουν την ISIS, τον, ε, το Ισλαμικό κράτος εναντίον των Πεσμεργά ή άλλων δυνάμεων στο Ιράκ και τη Συρία. Σίγουρα όμως ο αριθμό των μαχητών έχει αυξηθεί γιατί όλο και περισσότερο όταν έχουν ε, κατακτήσει έδαφος και περισσότερη χρηματοδότηση μπορούν να στρατολογήσουν περισσότερο κόσμο και να τους πιθαναγκάσουν ή να τους παραπλανήσουν για να γίνουν τμήμα του στρατού Υπάρχουν ακόμα και πολλοί οι οποίοι έρχονται από όλες τις άκρες του κόσμου για να συμμετάσχουν στον Ισλαμικό, στο Ισλαμικό κράτος στην ISIS. Δεν έχει μειωθεί λοιπόν η στρατιωτική δύναμη της ISIS, αντίθετα βλέπουμε μια αύξηση του αριθμού τους. Ξέρουμε βέβαια επί τόπου τη γεωγραφία του Κουρδιστάν, αλλά ξέρουμε επίσης ότι το ίσις ελέγχει μεγάλο τμήμα του εδάφους αυτού. Και οι πεσμεργά μπορούν να πολεμήσουν σε ορισμένες μόνο περιοχές. Το Σίντζαρ παραμένει προτεραιότητα και σκοπεύουμε να το απελευθερώσουμε και αυτό αλλά για άλλα τμήματα της χώρας υπάρχει ένα πολιτικά ευαίσθητο θέμα που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Αν το Κουρδιστάν ξεπεράσει τα εδάφη που θεωρούνται παραδοσιακά ως κουρδικά μπορεί να μην ε, γίνει δεκτό ευμενός από τους εκεί πληθυσμούς, αραβικούς πληθυσμούς και θα είναι πολύ δύσκολο για τους Πεσμεργκά να καταλάβουν εδάφη που δεν θεωρούνται παραδοσιακά Κουρδιστά. Θα θεωρήσουν δηλαδή ότι θέλουμε να καταλάβουμε και εδάφη πέραν των δικών μας. Ενώ δεν θέλουμε. Θέλουμε να ανακαταλάβουμε όλο το Κουρδιστάν αλλά με τα χαρά θα δεχόμασταν να είμαστε απλώς μέλος μια, ενός ευρύτερου συνασπισμού κατά του ίσης. Και θα ήθελα να το τονίσω αυτό οι χερσαίες δυνάμεις θα κερδίσουν τον αγώνα, οι αεροπορικές οι, μας βοηθάνε, τους ευχαριστούμε πολύ τους συμμάχους για όλα όσα έχουν κάνει για μας και τους βομβαρδισμούς, αλλά δεν θα κερδίσουν αυτοί τον πόλεμο. Πρέπει να υπάρξουν χερσαίες δυνάμεις και μέχρι τώρα μόνο η Πεσμεργά είναι η δύναμη που μπορεί να νικήσει το ίσις και να ανακτήσει γέες. Χρειάζεται λοιπόν πολύ περισσότερο, χρειάζονται πολύ περισσότερες χερσαίες δυνάμεις, ιδίως στη Συρία, και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα αφήσουμε κανένα μέρος στο ίσις για να μπορέσει να αναδιπλωθεί και να αναδιοργανωθεί και να επιστρέψει και να μας ξαναπολεμήσει. Δεν πρέπει να δοθεί, να αφαιθεί καθόλου χώρος για το ίσις ώστε να αισθανθεί ασφαλές. Για την εκπαίδευση, ναι, χρειαζόμαστε και εκπαίδευση γιατί αφού χρειαζόμαστε πολύπλοκα και προθυμένα όπλα και μας λένε ήδη «Ε, δεν έχετε τη γνώση για τη χρήση αυτών των όπλων πώς θα τα χρησιμοποιήσετε σωστό αλλά μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε από σήμερα ώστε να είναι έτοιμοι για να πολεμήσουν σε έξι μήνες από τώρα ας πούμε με αυτά τα πολύπλοκα και προθυμένα όπλα εάν μας τα δώσετε. Αν συνεχίσετε να μας λέτε δεν σας δώσουμε αυτά τα όπλα γιατί δεν έχετε ειδικού για να τα χρησιμοποιήσετε, ε, τότε πότε θα τους αποκτήσουμε. Πρέπει κάποτε να αρχίσουμε να τους εκπαιδεύουμε. Βοηθήστε μας να τους εκπαιδεύσουμε ώστε να είναι έτοιμοι οι μαχητές μας να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα πολύπλοκα και μοντέρνα όπλα. Εφόσον μάλιστα είμαστε και η πιο επιτυχής δύναμη που καταπολεμεί το ίσως αυτή τη στιγμή. Δεν θα είχε νόημα να, δώσουμε, να δώσετε όπλα σε εκείνους που δεν καταπολεμούν το ίσις όπως οι Πεσμεργά και να μην δίνετε προωθημένα όπλα στους Πεσμεργά που το κάνουν. Ναι, χρειάζεται και άλλη εκπαίδευση και στήριξη από εσά, χρειαζόμαστε μοντέρνα όπλα και τη γνώση του πώς χρησιμοποιούνται. Για τις ειρηνευτικές διαδικασίες μεταξύ ΠΚΚ και Τουρκίας. Πολλοί μίλησαν γι' αυτό. Εμείς πάντα λέγαμε ότι στηρίζουμε την ειρηνευτική διαδικασία στην Τουρκία. Πιστεύουμε δηλαδή ότι πρέπει ειρηνικά να διηθεί το πρόβλημα και να τύχει διαπραγμάτευσης. Αλλά δεν θα έπρεπε τίποτε να αλλάξει, να στρεβλώσει τις προσπάθειες αυτές με τρόπο άλλο εκτός από ειρηνικό. Υποστηρίζουμε λοιπόν τις διαπραγματεύσεις, τις συνομιλίες, τις διαπραγματεύσεις, ειρηνικές διαπραγματεύσεις και ελπίζουμε και οι δύο πλευρές να αναλάβουν να παίξουν ρόλο σε αυτή τη διαδικασία για να έχουμε αποτελέσματα. Επίσης υποστηρίζουμε οποιαδήποτε βοήθεια για θέλει οποιοδήποτε να χορηγήσει για να καταπολεμηθεί το ίσις. Στο κομμάνι αδέλφια μας που πολέμησαν κατά του ίσις πρέπει να στηριχθούν, τους αξίζει να στηριχθούν από τη διεθνή κοινότητα όσο και η Πεσμεργά σε άλλα τμήματα του Κουρδιστάν. Επίσης υπήρχε ένα ερώτημα για το Ιράν. Από την αρχή πρέπει να πούμε ότι οι Ιρανοί βοήθησαν μας βοήθησαν στην καταπολέμηση του ίσης από την αρχή και έχουν και αυτή η επιρροή στη, στο Ιράκ, ιδίως στη Βαγδάτη αλλά οποιαδήποτε συμμαχία κατά του ίσης νομι... Ε, ε, η συμμαχία κατά του ε, είναι κάτι το οποίο θα το εκτιμούσαμε. Άλλο θέμα για το καθεστώς του Άσαντ. Πολύ ενδιαφέρον. Πιστεύουμε ότι και το Ίσης και το καθεστώς Άσαντ έχουν αλληλοβοηθηθεί. Η διεθνής κοινότητα ζητούσε την απομάκρυνση του Άσαντ. Η μόνη πιθανότητα λοιπόν που είχε το καθεστώς αυτός ήταν να μπερδέψει τα πράγματα για να μην ξέρει η διεθνής κοινότητα ποια πλευρά να υποστηρίξει. Ώστε ο καθένας να σκεφτεί και να πει ποια πλευρά πρέπει να υποστηρίξω. Στην αρχή ήταν σαφές ποια πλευρά ήταν υπεύθυνη για την αιματοχυσία, αλλά δεν στηρίχθηκε επαρκώς η μετριοπαθής αντιπολίτευση στη Συρία. Το θέμα όμως αυτή τη στιγμή ακριβώς παραμένει, ήταν και είναι ακριβώς η στήριξη αυτής της μετριοπαθούς αντιπολίτευσης. Ούτε το καθεστώς Άσαντ ούτε το Ίσης αν εκμεταλλευτούν και οι δύο αυτή την έλλειψη υποστήριξης τη διεθνούς κοινότητας, τότε η αντιπολίτευση στη Συρία ποτέ δεν θα μπορέσει να πετύχει ή να μεγαλώσει την επιρροή της. Το ίσως πάντοτε εκμεταλλευόταν το γεγονός ότι ήταν σε θέση να, να σιωπήσει και να νικήσει την μετριοπαθή αντιπολίτευση στη Συρία. Αλλά για να υπάρξει κάποτε δημοκρατία στη Συρία το ίσις πρέπει να ιτηθεί. Όταν ιτηθεί το ίσις τότε ο λαός της Συρίας θα μπορέσει να έχει μια σωστότερη, καλύτερη επιλογή και η διεθνής κοινότητα θα μπορεί να τον στηρίξει πιο εύκολα. Για τη χρηματοδότηση τώρα. Το ίσις στηρίζεται από την πώληση πετρελαίου από τα δηληστήρια που κατέλαβε καθώς και από λίτρα που παίρνει από κόσμο που απάγει, από φορολόγησή του και επίσης από όλες τις περιοχές που έχει καταλάβει πουλάει τα δημητριακά, τη σοδιά και τα βιοτεχνικά προϊόντα για να πάψει αυτή η χρηματική υποστήριξη πρέπει ο κόσμος να μπορέσει να σταματήσει τη ροή και ιδίως τις δωρεές που δίνονται να παγώσουν δηλαδή ορισμένοι από τους λογαριασμούς που στηρίζουν το ίσις και οι διεθνείς τζιχαδιστές που έρχονται από διάφορα μέρη του κόσμου στη Συρία και μπαίνουν στο ίσις πρέπει να πιεστούν πολύ περισσότερο οι χώρες προέλευσής τους δηλαδή να διασφαλίσουν ότι δεν θα μπορούν τέτοιοι άνθρωποι να ε, ταξιδέψουν στο εξωτερικό για να πάνε να μπουν στο ίσις να ενταχθούν. Υπάρχουν χώρες που δεν έκαναν τίποτε για να τους σταματήσουν. Είναι και τα δύο σημαντικά λοιπόν, εκτός από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του να σταματήσει η ενδυνάμωσή του με διεθνείς τζεχαδιστές και με οικονομική στήριξη. Νομίζω ότι αυτά είναι τα κυριότερα ερωτήματα. Και τώρα κι άλλος γύρος. Αλλά... Λόγω του εισέλιψης χρόνου θα δώσω μονάχα ένα χρόνο <clears throat> στον στους ομιλητές και πρέπει να κλείσει ο κατάλογος των ομιλητών γιατί δεν θα έχουμε αρκετό χρόνο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Μπατσάνη για τις πληροφορίες που μας δώσατε σε σχέση με την ανησυχητική κατάσταση στην περιοχή του Κουρδιστάν και για τις ε, ε, ενέργειες του Ισλαμικού κράτους, του ISIS. Ένα από τα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν από τους ηγέτες των χριστιανών στο Ιράκ τους ε, το Ρίτς Λαφασά, τον ε, επικεφαλής των, χριστιανών ασυλοχαλδαίων. Η, τα χριστιανικά χωριά στο, στην πεδιάδα της Νινεβή έχουν ε, βρεθεί κάτω από απειλή. Είναι σημαντικά τα αγροκτήματα που έχουν εκεί οι χριστιανοί και οι ίσης όπως και το Κουρδιστάν βασίζονται σε αυτή την αγροτική παραγωγή για τις ανάγκες τους, ε, δεν έχει γίνει σπορά για την ε, επόμενη χρονιά και επομένω υπάρχουν πολλά μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία θα δημιουργηθούν για την επιβίωση του Ιρακινού Κουρδιστάν. Έχει κάθε λόγο λοιπόν το Ιρακινό Κουρδιστάν να απελευθερώσει το ταχύτερο δυνατόν αυτά τα χριστιανικά χωριά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν ποια είναι η άποψή σας για τις δυνατότητες να απελευθερωθούν αυτά τα χριστιανικά χωριά. Ευχαριστώ. Η Άννα Γκόμες. Ευχαριστώ κύριε Μπατζάνη. Θέλω να αποτίσω φόρο τιμή στους Πεσμεργά και τους ηγέτες τους για τον αγώνα που κάνουν εναντίον του Ισλαμικού κράτους στο Κομπάνι. Ξέρω ότι η κυβέρνηση του Ιρακινού Κουρδιστάν προσπαθεί να συλλέξει στοιχεία για τις μαζικές ε, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το ISIS και προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι θα υπάρξει και η αναγνώριση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την δίκη αυτών των υπευθύνων. Τι μπορείτε να μας πείτε σχετικά. Επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, ένα μέρος της επιτυχίας του ISIS για να μπορέσει να έχει μια ε, ισχυρή θέση στο Ιράκ οφείλεται και στην ε, δυσλειτουργία της Ιρακινής κυβέρνησης στην οποία συμμετέχετε κι εσείς. Βλέπετε λοιπόν να υπάρχει καλύτερη διακυβέρνηση στο Ιράκ και υπάρχουν καλύτερες προϋποθέσεις ώστε να μην ενισχύεται ο σεκταρισμός στο Ιράκ και πώς Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να σας βοηθήσει, περιορίστε μονάχα στην Βαγδάτη ή μπορεί να σας ενισχύσει και στην περιοχή του Ιρανικού, Ιρακινού Κουρδιστάν για να ενισχύσετε τις ικανότητές σας. Συναντηθήκαμε νωρίτερα κύριε Μπαρζάνη. Είμαι ο νέος πρόεδρος της Διακοινοβουλευτικής με το Ιράκ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την αποφασιστικότητα και το θάρρος που επιδεικνύουν οι μαχητές σας εναντίον του Ίσης. Από τις ε, τρεις προτεραιότητες που είπαμε στην αντιπροσωπεία, βασική βέβαια είναι όπως είπατε η καταστροφή του Ισλαμικού κράτους και η στήριξη επίσης ε, της Ιρακινής κυβέρνησης και η αποκατάσταση της κεραιότητας του Ιράκ. Πώς μπορούμε εμείς σαν αντιπροσωπεία να σας βοηθήσουμε πιο συγκεκριμένα σε επίπεδο στρατιωτικό και διπλωματικό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μπαρζάνη για την Τουρκία. Η Τουρκία ήταν φίλη του Ασάντ, μετά σταμάτησε να είναι φίλη του Ασάντ. Η Τουρκία προσπάθησε να συμφωνήσει με το ΠΚΚ, απ' την άλλη τώρα δεν προσπαθεί από ό,τι φαίνεται. Ε, στην αρχή σας εμπόδιζε να πάτε στο κομπάνι, τώρα σας επιτρέπει να πάτε στο κομπάνι. Ε, τι ακριβώς κάνει η Τουρκία. Σας διευκολύνει, σας εμποδίζει και τι μπορούμε να κάνουμε για να ακολουθήσει η Τουρκία τη σωστή οδό. Κύριος Χατζηγεωργίου. Διερωτώ με, εδώ και καιρό, γιατί το Ισλαμικό κράτος κατάφερε να προχωρήσει με τέτοια ταχύτητα προς το εμπρός. Μία εξήγηση είναι τα όπλα τους. Από την άλλη, έχω την αίσθηση ότι δεν θα μπορούσαν να προχωρήσουν με τόσο γρήγορο τρόπο αν δεν είχαν τύχη λαϊκή στήριξης. Θα ήθελα την ανάλυση σας. Ε, στηρίχθηκαν και γιατί από τους πληθυσμούς. Δεύτερον, για την Τουρκία. Ε, ποια είναι τα πραγματικά κίνητρα που ε, οδηγούν την Τουρκία στο να διστάζει να είναι πιο παραγωγική. Και τρίτον για το ΠΚΚ. Μήπως πρέπει να αποσυρθεί από την τρομοκρατική λίστα το ΠΚΚ. Σας ευχαριστώ. Μάτε τα ακουστικά σας παρακαλώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχήν για τις πληροφορίες που μας έχετε δώσει. Έχω δύο ερωτήματα τα οποία θα σας θέσω. Το πρώτο ερώτημα αφορά το δημοψήφισμα και η Ρόζαβα, το δυτικό Κουρδιστάν της Συρίας, έχει διακήρυξει την ανεξαρτησία του και κατανοώ την έννοια ενό δημοψήφισματος Οι Κούρδοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν για το δικό τους μέλλον. Το ερώτημα μου όμω είναι το εξή. Θεωρείτε ότι είναι δυνατόν να διατηρηθεί το Ιράκ σαν ένα ενωμένο κράτος και το ίδιο και η Συρία. Μπορεί να διατηρηθεί η συνοχή τους ή είναι αυτό ένα εμπόδιο για την ειρηνευσή στη Μέση Ανατολή. Δεύτερο ερώτημα. Το απεμπλουτισμένο ουράνιο το οποίο μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιείται σε αυτό τον πόλεμο και στο μέλλον. Γνωρίζετε ότι το, η χρήση του απεμπλουτισμένου ουρανίου έχει πολύ οδυνηρές συνέπειες για τους άμαχους, το είδαμε και στον προηγούμενο πόλεμο του Ιράκ και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στην ημέρα ιδιαίτερα της Γενικής Συνέλευσης. Τι, μπορεί, τι μπορείτε να μας πείτε σχετικά. Ο πρόεδρος δεν λέει σε ποιον δίνει το λόγο. Τουλάχιστον όχι στο μικρόφωνο. Την επόμενη εβδομάδα θα πάω στη Συρία και μπορεί να συναντηθώ και με τον Ασάντα. Τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω το Κουρδιστάν. Yes. Thank you, Chairman. Mr. Bazani. Κύριος Μαυρίδης, First, uh, Θα ήθελα καταρχάς να σας καλωσορίσω και εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω το θαυμασμό μου για τη μάχη που δίνεται για την ανεξαρτησία και την ελευθερία. Δύο σύντομες ερωτήσεις. Εδώ και λίγες εβδομάδες, εδώ στις Βρυξέλλες, στη θέση που είσαστε εσείς, είχαμε τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας. Δημόσια παραδέχθηκε ότι η Τουρκία είχε κάνει μια συμφωνία με το Ισλαμικό κράτος, το τρομοκρατικό Ισλαμικό κράτος για την ανταλλαγή των ομήρων. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι δυτικές χώρες ε, αρνούνται ότι έχουν επαφές με την τρομοκρατία και πληρώνουν υψηλό τίμημα γι' αυτό. Θα ήθελα το σχόλιο σας γι' αυτό και ένα δεύτερο μικρό σχόλιο τώρα εδώ. Αναφερθήκατε στα σύνορα αυτού που ονομάζεται Κουρδιστάν, στα όρια να το πω. Θεωρείτε ότι το Διαμπεκύρ και η περιοχή γύρω από το Διαμπεκύρ ανήκει στο κουρδικό κράτος. Uh, Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπαρζάνη, ή ο κύριο Σκάν τον ευχαριστούμε για τις ολοκληρωμένες πληροφορίες που έδωσε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο λαός του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως είπατε ο αγώνας αυτός να θεωρηθεί σαν ένας παγκόσμιος αγώνας εναντίον του ίσης, ε, του Ισλαμικού κράτους και όχι του μουσουλμανικού κόσμου λέτε ότι καταπολεμάτε την τρομοκρατία για πάνω από 100 χρόνια. Πώς βλέπετε να καταλήγει η προσπάθεια αυτή του κουρδικού λαού. Δεύτερη ερώτηση. Πόσο σημαντικό είναι έτσι ώστε να εμπλακούν οι τοπικές κυβερνήσεις, οι γειτονικέ κυβερνήσεις στον αγώνα εναντίον του ίσης και τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να εμποδίζει να πηγαίνουν να σειραίουν εκεί α, πολίτες από τον υπόλοιπο κόσμο υπέρ του Ισλαμικού κράτους. Πόσο χρειάζεται νομίζετε για να ολοκληρωθούν οι εχθροπραξίες, να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Αναφερθήκατε σε 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες. Ε, τι βοήθεια χρειάζεστε για να μπορέσετε να βοηθήσετε και εσείς τους πρόσφυγες αυτούς. Thank Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> κύριε Μπατζάνη, λέει ο κύριος Μποστινάρη, Μποστινάρου, θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για, τον, ε, για το σαφές και πραγματιστικό μήνυμα που δίνετε στην Επιτροπή μας. Είναι καιρό η Ευρώπη να σπάσει τα ταμπού και τις ουτοπικές σκέψεις που μας έχουν οδηγήσει στην κρίση που αντιμετωπίζουμε τώρα στη Μέση Ανατολή. Είναι φανερό ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αναθεωρήσει τη στρατηγική της, αν έχει βέβαια κάποια στρατηγική και όπως λέτε η Ευρώπη πρέπει να έχει μια νέα στρατηγική για την περιοχή αυτή που να είναι συνεκτική. Δεύτερον, αναφερθήκατε στο ρόλο της Συρίας και του Ιράν για τον αγώνα κατά του Ισλαμικού κράτους του ISIS. Πώς βλέπετε όμως το μέλλον του κουρδικού λαού στην περιοχή αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του προβλήματος αυτού και το γεγονός ότι εμπλέκονται τέσσερα κράτη στην περιοχή αυτή. Ποια είναι η δική σας αξιολόγηση για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπαρζάνη για το δύσκολο αυτό θέμα που μας έχετε δείξει και παρουσιάσει. Έρχομαι τώρα στο θέμα της Κομπάνη, όπου υπάρχει η μάχη αυτή η οποία συνεχίζεται για πάρα πολύ καιρό. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς 140 πεσμεργά, αν αυτός είναι ο σωστός αριθμός, θα μπορούσαν να αλλάξουν, να γίνουν την πλάστικα προς μια άλλη πλευρά και δεν θα είναι απλώς θύματα του εχθρού στο κομπάνι. Έχουν ζητήσει ε, Ορισμένοι ακόμα το λόγο. Ίσως λιγότερο από ένα λεπτό. Ο κύριος Σαφχάουζεν δεν έχει, φύγει. Η κυρία Σακορά θα έχει το λόγο. Κύριε Πασανή, θα ήθελα να σας δηλώσω το σεβασμό μου προς τον κουρδικό λαό και για τον αγώνα που δίνει για την επιβίωσή του και θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι για πρώτη φορά ίσως είναι ενωμένο περισσότερο παραποτέ. Στο παρελθόν και εσείς αλλά και μέλη της κυβέρνησης του Ιρακινού Κουρδιστάν έχετε ταχθεί υπέρ της ανεξαρτητοποίησης λέγοντας ότι αποτελεί το δικαίωμα του κουρδικού λαού ε, να αποκτήσει την ανεξαρτησία του. Θα ήθελα να μάθω αν είστε ακόμα υπέρμαχος αυτής της άποψης και αν ναι με ποιες όρους και ποιες προϋποθέσεις. Και δεύτερον, πριν από λίγους μήνες, η Βαγδάτη διέκοψε κάθε χρηματοδότηση προς το Αρμπίλ, κατηγορώντας το ότι κλέβει το πετρέλαιο που ανήκει σε όλους τους Ιρακινούς. Η διακοπή αυτής της χρηματοδότησης δημιούργησε πολύ μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας, με συνέπεια να μην υπάρχει δυνατότητα να πληρωθούν ακόμα και οι δημόσιοι υπάλληλοι και λαμβάνοντας υπόψη την πρωτοβουλία σας να αξιοποιείτε τη ζωτική σημασία για την κοινωνία πετρελαϊκές πηγές του Κουρδιστάν, θα ήθελα να μας πείτε τι συμφωνίες έχουν γίνει, έχουν υπογραφεί και με ποιους για την παραγωγή και εκμετάλλευση των πετρελοπηγών του Αρμπίλης. Ευχαριστώ. Πάρα πολλά ερωτήματα. Θα προσπαθήσω να είμαι συγκεκριμένο και σύντομο. Αλλά κάποια από τα ερωτήματα αυτά χρειάζονται πιο μακροσκελείς απαντήσεις. Για τα χωριά και τις πόλεις που είναι υπό τον έλεγχο του Ισλαμικού κράτους ακόμα. Κάποια από αυτά έχουν ήδη ε, απελευθερωθεί από το Άσο και μια άλλη πόλη, το Μπασίκα, θα μπορούσε να απελευθερωθεί σύντομα. Κάποια άλλα μέρη από το Κελεύ και το Καρακούς και άλλα μικρότερα χωριά που είναι πολύ κοντά στη Μοσούλη, γι' αυτό είναι δύσκολο να εξασφαλίσουμε την απελευθέρωσή τους, αλλά και να επιτρέψουμε στον πληθυσμό να επανέλθει, γιατί ανα πάσα στιγμή μπορούν να βρίσκονται μέσα στο βεληνικές πυροβολικού που μπορεί να ε, χρησιμοποιήσει το Ισλαμικό κράτος από τη Μοσούλη. Επομένως δεν είναι λογικό να περιμένει κανείς ότι θα γυρίσει αυτός ο πληθυσμός στα, στις αιστείες του εάν δεν απελευθερωθεί πλήρως η Μοσούλη από το Ισλαμικό κράτος. Μπορούμε λοιπόν να απελευθερώσουμε αυτά τα χωριά αλλά δεν θα γυρίσει ο άμαχος πληθυσμός γιατί θα είναι πάντα σε κίνδυνο επίθεσης από όλμους και από πυροβολικό του Ισλαμικού κράτους και θα επιτρέψει στον κόσμο αυτό να ζήσει σε αυτά τα μέρη. Πολλά λοιπόν θα εξαρτηθούν από μια ευρύτερη ενέργεια για την απελευθέρωση της Μοσούλης για να μπορέσουν να εξασφαλιστούν και οι κάτοικοι αυτών των περιοχών. Γιατί ήταν επιτυχής η ΆΕΣΙ στο Ισλαμικό κράτος. Αυτό ήταν ένα ερώτημα που θέσανε πολύ. Εγώ συμφωνώ ότι ο πόλεμος αυτός δεν είναι μονάχα το θέμα της ISIS. Ε, αντιμετωπίζουμε <clears throat> τις συνέπειες λανθασμένων πολιτικών που ακολούθηκαν στην Βαγράτη. Η ISIS είναι το αποτέλεσμα ενός μεγαλύτερου, ευρύτερου πολιτικού προβλήματος. Από τελέσματα αντιμετωπίζουμε και όχι ρίζες του προβλήματος. Αν η πολιτική κατάσταση στη Βαγδάτη είχε ένα περιεκτικό χαρακτήρα και συμπεριλάμβανε και τους Κούρδους και τους Σουνίτες και τους Σιήτες με έναν τρόπο ο οποίος ήταν ισοδίκαιος και δεν είχε πάρει σεκταριστικό χαρακτήρα. Δεν είχε τροποποιήσει το στρατό του Ιράκ από ένα εθνικό στρατό σε ένα σεκταριστικό στρατό. Πιστεύω ότι πάρα πολλοί δεν θα είχαν κανένα λόγο να υποστηρίξουν το Ισλαμικό κράτος, το ISIS εναντίον του Ιρακινού κράτους και δεν θα είχε καταρρεύσει ο Ιρακινός στρατός δεν θα είχε τύχει τέτοιας διαφθοράς και κατάπτωσης όπως έγινε στην πραγματικότητα, γιατί είναι φανερό ότι η προηγούμενη κυβέρνηση του Ιράκ δεν ήταν σε θέση να έχει ένα πραγματικό και επιτυχές πολιτικό σύστημα και να κρατήσει την ισχύ του στρατού. Θα έλεγα και πάλι ότι ο λόγος για την επιτυχία του Ισλαμικού, στρα... του Ισλαμικού κράτους, του ISIS, είναι γιατί πάρα πολλοί από τους ε, κατοίκους των σουνητικών περιοχών μπορεί να μην υποστήριζαν καθόλου το ΆΕΣΙΣ, αλλά το έπραξαν γιατί είχαν τόσο μίσος που έτρεφαν εναντίον του κεντρικού κράτους στη Βαγδάτη, ώστε να συμπλέψουμε οποιοδήποτε ο οποίος ήθελε να αγωνιστεί εναντίον της Βαγδάτης. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα και να επιληθεί, θα πρέπει να επιληθεί το πρόβλημα της διακυβέρνησης στη Βαγδάτη. Μπορούμε να κάνουμε στρατιωτικές επιχειρήσεις αλλά δεν θα, και να νικήσουμε τον εχθρό, αλλά αυτό δεν θα εξαλείψει το πρόβλημα. Αντίστοιχα προβλήματα θα υπάρξουν και στο μέλλον. Στο παρελθόν, πριν από την ISIS ήταν η Αλκάιδα, αύριο θα είναι κάποιος άλλος. Πρέπει να εξασφαλίσετε ότι τέτοιου είδους λανθασμένη συμπεριφορά και λανθασμένες πολιτικές δεν θα οδηγήσουν σε αντίστοιχα αποτελέσματα και δεν θα δημιουργηθούν και στο μέλλον οργανισμοί οι οποίοι θα στρέφουν τους ανθρώπους εναντίον των κυβερνήσεών τους. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο άμεσα. Πιστεύουμε ότι σε στρατιωτικό επίπεδο μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας υποστηρίξει με εξοπλισμό. Οικονομικά μπορούν να μας υποστηρίξουν σε οικονομικό επίπεδο να μας βοηθήσουν στρατιωτικά θέλουμε να υπάρξει άμεση σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Αρμπίλ, δηλαδή κουρδική συνιστόσα του Ιράκ. Δεν έχει νόημα να πρέπει να πηγαίνει ο εξοπλισμό στη Βαγδάτη να τον ελέγχουν και μετά, εάν το επιτρέψει η Ιρακίνη κυβέρνηση να έρθει στο Κουρδιστάν. Γιατί η Βαγδάτη θέλει να επιθεωρεί εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί εναντίον μια τρομοκρατικής οργάνωση τη στιγμή που μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει η Βαγδάτη να αντιμετωπίσει αυτόν τον τρομοκρατικό οργανισμό και βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε επίπεδο κατάρρευσης. Εμείς πολεμάμε και κερδίζουμε και θα πρέπει να πάρουμε τη βοήθεια και όχι να μας την αποστερεί η Βαγδάτη τη δυνατότητα να έχουμε άμεση παράδοση όπλων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε πολιτικό επίπεδο εμεί χρειαζόμαστε την υποστήριξη της Ευρώπης για το Ιρακινό Κουρδιστάν ως όαση σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή αυτή και ως στοιχείου ενίσχυσης της συνύπαρξης κοινωνιών και ομάδων από διαφορετική εθνοτική και θρησκευτική προέλευση. Χρειαζόμαστε λοιπόν την υποστήριξή σας για να μπορέσει το Κουρδιστάν να γίνει ένα ακόμα πιο επιτυχές υπόδειγμα στην Μέση Ανατολή, σε μια περιοχή γεμάτη με αβεβαιότητα και χάος. Η επιτυχία του Κουρδιστάν είναι κάτι το οποίο πρέπει να υποστηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να μας αφήσετε στην τύχη μας. Χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας και οικονομικά, γιατί πέραν των προβλημάτων που έχουμε με το δικό μας λαό, γιατί δεν παίρνουμε καμία χρηματοδότηση από τον εθνικό προπολογισμό. Όπως είπα έχουμε 1,5 εκατομμύρια εκτοπισμένους και πρόσφυγες από τη Συρία και από το Ιράκ και χωρίς την υποστήριξη σε οικονομικό επίπεδο το περιφερειακό κράτος του Κουρδιστάν δεν μπορεί να συνεχίσει να υποστηρίζει τα άτομα αυτά τη στιγμή που έρχεται ο χειμώνα και είναι όλο και πιο δύσκολο για τα άτομα αυτά να ζήσουν σε στατόπεδα προσφύγων κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Ελπίζω λοιπόν ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες της διεθνού κοινότητας και η χρηματοδότηση της διεθνού κοινότητας θα είναι πιο γενναιόδορη από ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής. Αυτά είναι λοιπόν τα τρία στοιχεία που θέλω να τονίσω. Χρειαζόμαστε στρατιωτική υποστήριξη, οικονομική υποστήριξη και πολιτική υποστήριξη και στους τρεις αυτούς τομείς πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή ε, υποστήριξη και ο ηγετικός ρόλος της Ευρώπη θα είναι πάρα πολύ σημαντικός. Τουρκία, δεν μπορώ τώρα να μιλήσω εξ ονόματος της Τουρκίας. Έχουν τις δικές τους πολιτικές. Η Τουρκία είναι γείτονά μα. Μπορεί να διαφωνούμε με πολλές από τις πολιτικές τους, από ό,τι κατανοούμε, από ό,τι έχουμε μάθει από αυτούς. Δεν μπορούν να δώσουν την υποστήριξη που ζητήσαμε λόγω της κατάστασης ομοιρίας των διπλωματών τους και επειδή τότε λάμβαναν χώρα οι προεδρικές εκλογές. Τώρα όλα αυτά έχουν περάσει και ελπίζουμε ότι η Τουρκία θα αναλάβει δράση και θα υποστηρίξει πολύ περισσότερο τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Πέραν αυτού βέβαια δεν μπορώ να πω τίποτα, εναπόκειται στην Τουρκία να εξηγήσει τη στάση της. Κατά πόσον τώρα θα πρέπει να τροποποιηθεί το καθεστώς του ΠΚΚ και να μην χαρακτηρίζεται πια ως τρομοκρατική οργάνωση. Εμείς ποτέ δεν θεωρούσαμε το ΠΚΚ ότι είναι τρομοκρατική οργάνωση. Γι' αυτό φυσικά δεν υποστηρίζουμε το να μείνει το ΠΚΚ ως τρομοκρατική οργάνωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση για το δημοψήφισμα. Αν θα κρατήσει ενωμένη τη χώρα μας το δημοψήφισμα. Α είμαι σαφή και όχι διπλωματικό. Αν δείτε την ιστορία του Ιράκ, το Ιράκ δεν ήταν ποτέ σταθερό και ειρηνικό. Ούτε στο εσωτερικό του, ούτε και εναντί των γειτονικών χωρών. Το να επιμείνουμε στο να κάνουμε συνέχεια τα ίδια σφάλματα θα οδηγήσει πάντα στα ίδια αρνητικά αποτελέσματα. Το Ιράκ πλήττεται από την έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των Σουνιτών, των Σιητών και των Κούρδων. Δεν υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη. Πρέπει να βρεθεί ένα κοινό έδαφος για να μπορέσουν αυτοί οι λαοί να ζήσουν μαζί σε μια χώρα. Και αυτό δεν θα γίνει εάν δεν υπάρχουν επαρκείς εγγύησεις ότι καμία από αυτές τις κοινότητες δεν θα είναι κυριαρχούμενη από τις άλλες κοινότητες. Αν δείτε την ιστορία των Κούρδων, εμείς έχουμε υποστεί χημικούς βιομηχανισμούς. Έχουμε αντιμετωπίσει φόνους, βασανιστήρια, εκτοπίσεις. Όλα αυτά είναι πολύ νοπά στη μνήμη μας. Πώς μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στο μέλλον του λαού μας, αν δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι όλες αυτές οι ομότητες δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον. Ο φεδραλισμός δυστυχώ ούτε και αυτό έδωσε τι απαραίτητε εγγύησει, γιατί η κυβέρνηση τη Βαγράτης δεν εφάρμοσε ένα ομοσπονδιακό επίπεδο. Μια συνομοσπονδία μπορεί να είναι μια λύση, γιατί οι Κούρδοι και οι άλλες συνιστώσεις του Ιράκ θα πρέπει να νιώθουν ασφάλεια, θα πρέπει να ξέρουν ότι το μέλλον τους θα είναι ασφαλές και το μέλλον των παιδιών τους θα είναι ασφαλές. Έχουμε άλλα πέντε λεφτά. Κάποιος από εσάς είπε ότι θα πάει στη Συρία να συναντήσει τον κύριο Μπασάρα Λασάδ. Νομίζω ότι ένα ερώτημα μπορεί να θέσει και αυτό φτάνει. Να το ρωτήσει γιατί οι Κούρδοι δεν αποτελούν ούτε και τώρα πολίτες της Συρίας. Είναι εδώ και αιώνες στη Συρία. Ζούνε στις περιοχές του Κουρδιστάν που ανήκουν στη Συρία. Γιατί δεν αναγνωρίζονται όμως ακόμα ως ίσοι πολίτες της Συρίας αν θέλουν να έχουν την υποστήριξη των Κούρδων, το καθεστώς της Συρίας θα πρέπει να αντιμετωπίσει τους Σύριους ε, Κούρδους ως ίσους πολίτες με τους υπόλοιπους πολίτες της Συρίας. Ευχαριστώ, λέει και ο θέσα το ερώτημα. Αν πιστεύουμε ότι το Κουρδιστάν είναι, ε, περιλαμβάνει τη Βόρεια Συρία. Αν λάβετε υπόψη το πόσο μεγάλο είναι το Κουρδιστάν μαζί με, τη, με τους Κούρδους της Συρίας, ε, του Ιράν και της Τουρκίας, είναι μια μεγάλη περιοχή η οποία έχει διαιρεθεί μετά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο σε τμήματα. Έχουμε όμως μια πραγματικότητα που έχει διασπασμένο Κουρδιστάν, το Ιρακινό Κουρδιστάν, το Τουρκικό Κουρδιστάν, το Συριακό και το Ιρανικό. Εμείς λοιπόν εστιάζουμε την προσοχή μας σε αυτά που γίνονται στο Ιράκ. Ξέρουμε πόσο ευαίσθητο είναι το θέμα αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι κάθε περιοχή έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δεν θέλουμε να επισέλθουμε στα εσωτερικά οποιασδήποτε χώρας, αλλά υποστηρίζουμε πάντα την ιδέα ότι οι Κούρδοι που ζουν σε αυτές τις χώρες θα πρέπει να αποφασίσουν μόνοι τους το μέλλον που θα θέλουν να έχουν και τη σχέση που θα πρέπει να έχουν. Αν λοιπόν οι Κούρδοι της ε, Συρίας και δεν εκπροσωπούν όλους τους Κούρδους της Συρίας, υπάρχουν πολλοί άλλοι πέραν αυτών που εκπροσωπούνται από το YPG, Οτιδήποτε σύστημα λοιπόν επιλέξουν, εμείς θα το υποστηρίξουμε και ελπίζουμε ότι και εσείς θα το υποστηρίξετε. Θα υποστηρίξετε τα αιτήματα των Κούρδων όπου και αν βρίσκονται. Okay, well, I don't know if uh, In terms of, there was a question about how many υπήρξε ένα ερώτημα για το οι πεσμαλικά πήγαν στο κομπάνι. Αυτό σας το λέω για να είναι σαφές. Ήμασταν <clears throat> έτοιμοι να στείλουμε περισσότερους. Αλλά επί τη βάση των ετοιμάτων των αγωνιστών που υπερασπίζονται το κομπάνι, μας είπανε ότι δεν θέλουμε μία μάχημη δύναμη, θέλουμε απλώς ειδικού για να χρησιμοποιήσουν το πυροβολικό. Επομένως ο αριθμός των Πεσμέργα βασίστηκε στις ανάγκες και τις αιτήσει που ήταν από τους υπερασπιστές του κομπάνι και μόνο. Αλλιώς ήμασταν έτοιμοι και είμαστε ακόμα έτοιμοι να στείλουμε περισσότερους μαχητές στο κομπάνι. Αν η ανεξαρτησία τώρα είναι στόχος ή όχι. Κοιτάξτε, είναι ένα θεόπεμπτο δικαίωμα των Κούρδων όπως και ουδήποτε άλλου λαού στον κόσμο. Ό,τι είναι λοιπόν καλό για τους άλλους είναι καλό και για τους Κούρδους. Αν κάποιοι θέλουν να εκχωρήσουν την ανεξαρτησία τους, ε, ε, τότε αυτό δεν θα εντυπωσίαζε μάλλον πολύ κόσμο αλλά νομίζω ότι αν θεωρείται η ανεξαρτησία θετικό πράγμα σε όλο τον κόσμο, αυτό θα πρέπει να ισχύει και για τους Κούρδους. Πρέπει ισότιμα και ελεύθερα να ζουν με αρμονία και ειρήνη, γιατί το αξίζουν όπως και όλοι οι λαοί του κόσμου. Καταλαβαίνουμε την πραγματικότητα, καταλαβαίνουμε τις ευαισθησίες. Δεν θέλουμε να δημιουργούμε προβλήματα και γι' αυτό θέλουμε να ακούτε άμεσα τον λαό και τις ανάγκες του λαού μας και τι αξίζει στον λαό μας. Υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις αλλά νομίζω δεν έχουμε πια άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω ο κύριος Μπαρζανή ζητώ συγγνώμη για το ανάφησα κάποιες ερωτήσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Μπαρζανή για μια ακόμη φορά. I think uh, that uh, there's Νομίζω ότι πράγματι υπάρχει πολύ υποστήριξη, διάχυτη υποστήριξη στην υπόθεσή σας, στην περιοχή σας, στον λαό σας και οι άλλοι λαοί της περιοχής επίσης την χάνουν της υποστήριξής μας στα πλαίσια του κράτους δικαίου. Ελπίζω να βελτιωθούν τα πράγματα σύντομα θα παραμείνουμε σε επαφή. Ε, χαιρετίζω επίσης τους εκπροσώπους της γεζιδικής κοινότητας στη Γερμανία και τον Κιζιλάν και άλλους και σας εύχομαι σας μάλλον σας ε, Εύχομαι κάθε επιτυχία στο, στις προσπάθειές σας και σας δίνω τη δική μου υποστήριξη για τις δύσκολες στιγμές που περνάτε και σας ευχαριστώ που ήρθατε στη συνεδρίασή μας. Κλείνει το σημείο αυτό της ημερησίας διάταξης και περνάμε στο επόμενο σημείο που έχει να κάνει με τις εκλογές στην Τινησία. Είναι μεγάλη σημασία σε αυτές οι εκλογές που έλαβαν χώρα στην Τινησία γιατί κατέδειξαν ότι μπορούν να υπάρξουν λύσεις που ανοίγουν δρόμους για το μέλλον και πιστεύω ότι και εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο, ιδίως οι Γάλλοι φίλοι μας και ο συνδυασμός της πολιτικής, κοινωνικής και πολιτικής εξέλιξης είναι εφικτός. Και αυτό μας είπαν οι εμπειρογνώμονες ότι αυτό είναι κάτι το εφικτό επειδή υπήρξε μια μέση τάξη στην ε, την Ισία. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν ιδιαίτερα και τον Μιχαελ Γκάλερ, ο οποίος αγωνίστηκε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία ως παρατηρητής από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και επίση θέλω να ευχαριστήσω όλου αυτού οι οποίοι υπό την ηγεσία του κυρίου Γκάλερ πήγανε στην Επιτροπή ε, Παρακολούθησης των Εκλογών. Μπορείτε να φύγετε παρακαλώ, κυρία Λέζιν. Κυρία Μήπως μπορείτε να φύγετε από την αίθουσα. Κοίτα. Και έπαιξε σημαντικό ρόλο ο κύριος Γκάλερ και η Επιτροπή μας ε, Παρακολούθηση επίσης και ο κύριος ε, Παντσέρη, ο οποίος είναι ο επικεφαλής αντιπρόσωπείας μα εκεί, ο Μίχαελ πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Υπήρξαμε παρατηρητές των εκλογών στο, στην Τίνιδα κατά τη διάρκεια των εκλογών της 26ης Οκτωβρίου ήταν παρόν και ο κύριος Παντσέρη, η κυρία Βαλενθιάνο, η κυρία Κριστίν Βερσιά, ο Ζόρντι Σεμπάστια, ο Φάμπιο Μάσιμο Καστάλτο, Νικόλα Μπαΐ. Μήπως μπορείτε να συνεχίσετε τη συζήτησή σας έξω, γιατί έχουμε ένα άλλο θέμα να συζητήσουμε εδώ. Τώρα μιλάμε για την Τινησία και όχι για το προηγούμενο θέμα, λέει ο κύριος Γκάλερ. Θα χαιρόμουν πολύ αν το εκτιμούσατε και εσείς. Αν δει στον αραβικό χώρο, είναι φανερό ότι ένα θετικό παράδειγμα ως η Ισία μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα. Μετά από τρία χρόνια έχουμε λοιπόν την πρώτη τέτοια περίπτωση εκλογών που έχουν λάβει στην ε, Τινησία Έχουν λοιπόν η τίνηση μέσα σε τρία χρόνια περατώσει και τη συνταγματική διαδικασία. Δεν έγιναν λοιπόν όλε οι προσπάθειές μας επιματέω. Έχει καταλήξει τελικά μια διαδικασία σε συνένεση που οδήγησε σε ένα σύγχρονο σύνταγμα, ένα σύνταγμα το οποίο ε, λαμβάνει υπόψη και τις αιτήσει της κοινωνίας των πολιτών και δημιουργεί ένα πλαίσιο, δημιουργήσε και το πλαίσιο με στο οποίο Μπόρεσαν να γίνουν εκλογές, εκλογές που δεν μποϊκοτάρισε καμία πολιτική δύναμη, αντίθετα όλες οι δυνάμεις που ήθελαν να συμμετάσχουν μπορέσαν να συμμετάσχουν και μπορέσαμε να διαπιστώσουμε <clears throat> ότι τόσο η προετοιμασία όσο και η διεξαγωγή των εκλογών έγιναν σύμφωνα με τους τεθειμένους κανόνες και εγώ είπα στον ε, τινησιακό τύπο ότι το πιο εντυπωσιακό με αυτές τις εκλογές είναι ότι δεν υπήρξε κανένα εντυπωσιακό γεγονός κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας. Αυτή η διαδικασία λοιπόν έγινε με τόσο ομαλό τρόπο όσο δεν θα μπορούσε κανείς να φαντιστεί. Έχουμε για πρώτη φορά, είχαμε για πρώτη φορά ένα ενιαίο κατάλογο ψηφοφόρων. Στο παρελθόν είχαμε αυτούς οι οποίοι είχαν εγγραφεί εθελοντικά και αυτούς οι οποίοι είχαν προκύψει από τις ληξιαρχικές καταστάσεις, κάτι το οποίο είχε οδηγήσει στο να έχουμε 4,3 εκλογές, εκλογής το 2011, ενώ αυτή τη φορά με τις προσπάθειες της Εκλογικής Επιτροπής ώστε να πείσει τους πολίτες να εγγραφούν εθελοντικά είχαμε ένα εκατομμύριο περίπου πρόσθετους εκλογής αλλά στο τέλος ψήφισαν μονάχα 3,1 εκατομμύρια. Δηλαδή περίπου τα 70% των εγγεγραμμένων ε, των ε, αυτών που θα μπορούσαν να εγγραφούν, εγγράφησαν. Αυτό δεν είναι ικανοποιητικό για μένα. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε και με τους ε, τινήσιους ομολόγους μας πώς θα μπορέσει να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών. Υπήρξε μια ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. 14.000 ε, παρατηρητές από διάφορους φορείς ήταν παρόντες στις εκλογές, περίπου χίλιοι διεθνείς παρατηρητές και η δική μας ε, αντιπροσωπεία παρακολούθησης ήταν η σημαντικότερη για τη μακροχρόνια παρακολούθηση των εκλογών. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξαν λοιπόν αντίστοιχες επιτροπές παρακολούθησης και από το Συμβούλιο της Ευρώπης με ε, συνεχή παρουσία στο χρόνο, με μεγάλη χρονική διάρκεια. Από την Αφρικανική Ένωση, από τις γαλλόφωνες χώρες υπήρξαν άλλες επιτροπές παρακολούθησης και νομίζω ότι έχουμε καταλήξει σε ένα θετικό αποτέλεσμα, όπως είπα προηγουμένως, για την εκλογική διαδικασία η οποία είχε άψογο χαρακτήρα και η ανεξάρτητη εκλογική ε, επιτροπή έκανε ένα σημαντικό και πάρα πολύ θετικό έργο. Τα αποτελέσματα των εκλογών σημαίνουν ότι το προηγούμενο κόμμα της εξουσίας είναι τώρα το δεύτερο ισχυρότερο κόμμα. Το μεγαλύτερο τώρα κόμμα είναι το Κοσμικό Κόμμα Νίντα Τούνης. Το κάλεσμα για την Τίνιδα, αν το πω στα γερμανικά, στην αντίστοιχη γλώσσα, κύριο Σέξι, μαζί με άλλους υποψηφίους θα πρέπει να διεκδικήσει την Προεδρία. Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και στις 28 Δεκεμβρίου θα προβλέπεται να γίνει ο επόμενος γύρος μετά τις 23 Νοεμβρίου. Είναι ενδιαφέρον τα τρία κόμματα της ε, κυβέρνησης, η λεγόμενη Τρόικα, υπέστησαν μια ε, απόρριψη σε μεγάλο βαθμό από τον πληθυσμό. Ένα κόμμα από αυτά τα τρία πήρε μοναχα τέσσερα, τέσσερις έδρες και το κόμμα του Τζάφα Μπακατόλ πήρε μοναχα μία έδρα στις εκλογές. Βλέπουμε λοιπόν μία εξέλιξη όπως είδαμε και στην κεντροανατολική Ευρώπη μετά από τις πρώτες ελεύθερες εκλογές όπου τα προηγούμενα κόμματα της εξουσίας τιμωρήθηκαν μέσα σε εισαγωγικά από τους εκλογείς. Αλλά το βασικό είναι ότι υπήρξε ευρεία αποδοχή των αποτελεσμάτων αυτής της εκλογικής διαδικασίας και η Επιτροπή Παρακολούθησής μας που ήταν εκεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου ήδη με την επικεφαλής την κυρία Άνεμι Νέιτς Ρίτενμπρουκ παρέμεινε και με, μέχρι το δεύτερο και θα μείνει μάλλον μέχρι το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών θα επανέλθει τον Ιανουάριο για να μας δώσει μια συνολική εικόνα. Αφού περατωθεί και ο τελευταίος γύρος των προεδρικών εκλογών, η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν και οι αντιπροσωπείες μας θα παραμείνουν σε επαφή με τις τοπικές πολιτικές δυνάμεις που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο και θα συνεχίσει και η υποστήριξη που δίδουμε για την περαιτέρω δημοκρατικοποίηση και η ομάδα αυτή για την υποστήριξη της δημοκρατίας. Α, ναι, δεν προεδρεύει πια ο Έλμαρ Μπρόκ, το ξέχασα. Αυτή λοιπόν η επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για την υποστήριξη των δημοκρατικών δυνάμεων εκεί. Ελπίζω ότι θα μπορέσει να συνεχιστεί και να περατωθεί όλη αυτή η διαδικασία και θέλω να ευχαριστήσω όσους συναδέλφους είναι ακόμα εδώ οι οποίοι έχουν λάβει μέρος σε αυτήν την ε, ε, Επιτροπή Παρακολούθησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Παντζέρη. Αλλά δεν είναι εδώ. Είναι στην αντιπροσωπεία με τις χώρες του Μαγκρέμπ. Θα σας δώσω το λόγο, περιμένετε. οι προεδρικές εκλογές της 23ης Νοεμβρίου και της 28ης του Δεκεμβρίου είναι θέματα τα οποία θα παρακολουθήσουμε και εν τω μεταξύ θα ανταλλάξουμε ε, θα έλεγα ιδέες και εμπειρίες από μια διαδικασία η οποία είναι ένα παράδειγμα ένα δημοκρατικό κράτος που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λοιπόν θα περάσουμε στην ανταλλαγή των απόψεων τώρα. Η κυρία Γκάμπριελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ τα μέλη της αντιπροσωπείας. Ευχαριστώ για όλη τους την εργασία και τα συμπεράσματά τους. Αρχίζω λέγοντας ότι μπορούμε πράγματι να εκφράσουμε τη χαρά μας για τα αποτελέσματα των εκλογών στην Τινησία που έγιναν ήρεμα, διαφανώς και με σεβασμό των εκλογικών νόμων που θεσπίστηκαν από την επανάσταση του Γιασεμνιού. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η έκκληση μπορεί να ακουστεί με τρεις τρόπους. Πρώτον, η καμπάνια που έγινε για να αυξηθεί ο αριθμός των εκλογέων κατά ένα περίπου εκατομμύριο από το 2011 είναι κάτι πολύ σημαντικό και σίγουρα προϊονίζει θετικά για το δημοκρατικό μέλλον της χώρας γιατί γράφτηκαν περισσότεροι νέοι και γυναίκες στους εκλογικούς καταλόγους χωρίς τους οποίους δεν μπορεί να είναι πλήρη μια πραγματική δημοκρατία. Σήμερα το ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί ακόμη η εκλογική συμμετοχή διότι υπάρχει σταθερή βάση και μπορούν επομένως αποδείχτηκε να υπάρχουν περισσότερες εκλογές από το 2011. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι αποδείχθηκε ότι μπορούν να υπάρξουν, μπόρεσαν να υπάρξουν μηχανισμοί πολύπλοκοι εκλογικών διαδικασιών σε πολύ λίγο χρόνο. Και αυτό είναι πολύ θετικό για ένα δημοκρατικό κράτος το οποίο θα είναι επιπλέον σε θέση, πλέον σε θέση να εφαρμόσει τις απαραίτητες οικονομικές και άλλες δομικές μεταρρυθμίσεις, κατά καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και η μείωση του, της ανεργίας σε, διάφο, σε ειδικές, ιδίως ορισμένες περιφέρειες της νησίας, είναι κάτι επίσης σημαντικό. Επίσης ο νόμος για την ισότητα ανδρών και γυναικών είναι επίσης κάτι θετικό αν και δεν σημειώθηκαν σημαντικές προόδια από το 2011. Πάντως το πεδίο εφαρμογής του έγινε πιο συγκεκριμένο και θα ήθελα να δούμε πώς θα μπορούσαν οι γυναίκες να συμμετάσχουν ακόμη περισσότερο στην πολιτική ζωή της Τινησίας και καταλήγω λέγοντας ότι πρόκειται για, για εκλογική διαδικασία πολύ ενθαρρυντική αν και δεν μπορούμε να πούμε ότι επιτεύχθηκαν όλα όσα θα θέλαμε ήδη. Πάντως μπορούμε στο εξή να υπολογίζουμε σε ένα πολιτικό σύστημα που αν και πρέπει ακόμη να αποδείξει ότι είναι σε θέση να λύσει τα προβλήματα παρόλα αυτά διαθέτει μια ισχυρή βάση και δεν πρέπει να πέσει σε έναν διπολισμό που θα εμποδίσει τις μεταρρυθμίσεις. Σας ευχαριστώ πάντως για την ε, αποστολή που χάρη στις παρατηρήσεις και τα αποτελέσματά της θα μπορέσει να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκαμπριέλ. Α, ο κύριος Παντσέρη είναι παρόν τώρα. Ζητώ συγγνώμη αλλά Είχαμε μια ακρόαση με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Είμαι εισηγητή για την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έπρεπε να είμαι εκεί. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο πάντως. Νομίζω ότι ο κύριος Γκάλα ήδη είπε πάρα πολλά πράγματα. Προφανώς κατήφθηνε τις εργασίες της αντιπροσωπείας μας με εξαιρετικό τρόπο. Είναι αλήθεια ότι οι εκλογές αυτές διεξήχθησαν με πολύ καλό τρόπο. Υπήρχαν ε, λιγότερες εντάσεις από ότι το 2011. Υπήρχαν ε, περισσότερες ε, θα έλεγα ικανότητες, υπήρχε μεγαλύτερη ηρεμία. και όπως είπα και η προεκλογική εκστρατεία γενικά εξελίχθηκε σε ένα κλίμα ειρηνικό. Όλοι μπόρεσαν να παρουσιάσουν ελεύθερα τα προγράμματά τους και σεβάστηκαν όλοι τους κανόνες της προεκλογικής εκστρατείας. Είμαι πεπισμένος ότι αυτές οι εκλογές είναι μια θετική στροφή για την χώρα. Και είναι επίσης σαφές ότι θα πρέπει να χαιρετήσουμε σαν εκλογικοί παρατηρητές τη διαδικασία. Δύο σημεία μόνον, σύντομα. Και τελειώνουμε αυτά. Η Τινησία μετά από την ψηφοφορία και μετά από τους δύο γύρους των προεδρικών θα έχει αντικειμενικά ολοκληρώσει την διαδικασία δημοκρατικής σταθεροποίησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρόκειται για μια μικρή χώρα μένα, αλλά μπορεί να είναι σημείο αναφοράς για την υπόλοιπη περιοχή και για την κοινή γνώμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι η κοινή γνώμη στην Ευρώπη στην αρχή είδε με εμπιστοσύνη την λεγόμενη Αραβική Άνοιξη, αλλά την εμπιστοσύνη αυτή διαδέχθηκε μια έλλειψη πικρίας. Ενώ η διαδικασία της Τίνιδος δείχνει ότι οι εξεγέρσεις αυτές είχαν νόημα, ότι υπάρχει μια κοινωνία η οποία μπορεί να ολοκληρώσει την δημοκρατική διαδικασία. Και αυτό θα επανεμπνεύσει θα έλεγα την ευρωπαϊκή κοινή Τέλος, μια επιπλέον παρατήρηση ίσως δεν είναι δική μου θα έλεγα. Δεν μπορούμε να ικανοποιηθούμε και να αρκεστούμε σε αυτά ε, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήγαν καλά οι εκλογές, σταθεροποιείται η χώρα, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να επαναφαθεί. Θα πρέπει οικονομικά να βοηθήσει τη χώρα. Υπάρχει μια οικονομική κρίση στην Τινησία, μια κοινωνική σαν συνέπεια της προηγούμενης και γι' αυτό θα πρέπει να συνοδεύσουμε τη διαδικασία δημοκρατικής σταθεροποίησης οικονομικά. Ευχαριστώ λοιπόν και τον Κάλε φυσικά ο οποίος ε, ηγήθηκε της αντιπροσωπείας, να ευχαριστήσω και όλους όσους πήραν μέρος στη διαδικασία εκλογικής παρατήρησης. Ευχαριστώ κύριε Παντζέρη. Ε, ε, δεν, δεν ήθελα απλά να πω ότι είχαμε κάθε συμφέρον να σας ακούσουμε. Σας ευχαριστώ. Δεν θέλω να, επανε, λάβω, λέει κυρία Βέρζη, αυτά που είπαν οι συνάδελφοί μου. Σύμφωνα απόλυτα με τους συναδέλφους, απλώς θέλω να σταθώ σε ορισμένα θέματα. Νομίζω ότι πράγματι η Τινησία έχει μπορέσει να περάσει ένα σημαντικό ορόσημο. Υπήρξε βέβαια περιορισμένος αριθμός ε, εγγεγραμμένων, θέλω να υπογραμμίσω όμω αυτό που είπε και η κυρία Γκαβριέλ, ότι οι νέοι ε, δεν ήταν αρκετά παρόντες στην εκλογική διαδικασία. Αυτό είναι ένα κακό μήνυμα και κακό ιονός και θα πρέπει να παρακολουθήσουμε καλύτερα τα θέματα αυτά. Σίγουρα είπανε πολλοί ότι ήταν υπερβολικά ήρεμες οι εκλογές και αυτό δείχνει την κατάσταση των πραγμάτων. Κυριάρχησαν τα δύο μεγάλα κόμματα στις ε, προεκλογικές ε, εκδηλώσεις και η συζήτηση είχε αρκετά διπολικό χαρακτήρα. Δεν αντιμετώπισε τα ουσιαστικά θέματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες της Τινησίας και αυτό εξηγεί σε κάποιο βαθμό την ε, συμμετοχή ή μάλλον τη μη συμμετοχή ορισμένων ε, στρωμάτων του πληθυσμού. Η όλη συζήτηση για τον κοσμικό κόσμο, για το κοσμικό ή θρησκευτικό ε, πλαίσιο της χώρας επέτρεψε να παρακαμφθεί το θέμα των οικονομικών προβλημάτων. Θέλω όμως να υπογραμμίσω το γεγονός ότι υπήρξε ένας σημαντικός ε, ρόλος των μέσων ενημέρωσης και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ευήκοοι σε αυτή την κατάσταση που έχει να κάνει με τα μέσα ενημέρωσης. Τα μέσα ενημέρωσης και η έλλειψη οικονομικής δυνατότητας έφεραν στην τρίτη θέση ένα κόμμα το οποίο θα μπορούσε να έχει καλύτερη θέση. Λοιπόν πρέπει να είμαστε επάγρυπνοι για όλα αυτά τα θέματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο μεγάλα κόμματα τα οποία κυριαρχούν πλήρως Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να έχει μια απόλυτη πλειοψηφία. Θα είναι δύσκολο να βρεθεί μια πλήρης πλειοψηφία. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις στήρες αντιπαραθέσεις αλλά πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για τα τεκτενόμενα στην ισία. Έχουμε και τις προεδρικές εκλογές στις 23 Νοεμβρίου. Είναι σημαντικές λοιπόν αυτές οι προεδρικές εκλογές και πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι κάποιες πολιτικές παρατάξεις δεν έχουν παρουσιάσει υποψηφίους. Αλλά δεν πρέπει να είμαι απεσιόδοξη. Πιστεύω ότι πράγματι η Τινησία είναι ένα θετικό παράδειγμα για όλη την περιοχή. Βρίσκεται στην φάση αυτή της δημοκρατικής μετάβασης. Μας το είπανε πάρα πολύ και νομίζω ότι αυτό εξηγεί πολλά. Πρέπει να στοιχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί σε σχέση με την Τινησία, σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο, σε σχέση με την ανάγκη μεταρρυθμίσεων, για τα μέσα ενημέρωσης, για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, για τις διεκδικήσεις της κοινωνίας των πολιτών. Πιστεύω λοιπόν ότι η κοινωνία των πολιτών είναι αρκετά καλά οργανωμένη στην ε, Ισία και αν έχει φτάσει σε αίσιο πέραση η συνταγματική διαδικασία, αυτό οφείλεται στην κοινωνία των πολιτών. Θα πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν να βασιζόμαστε στην κοινωνία των πολιτών, όντα επάγρυπνοι εμεί και προσπαθώντας να λάβουμε υπόψη το σύνολο των εμπλεκομένων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ απέραντα κύριε Πρόεδρε. Θέλω καταρχήν να ε, συγχαρώ όλους τους συναδέλφους που πήγαν στην Τινησία να παρατηρήσουν αυτές τις εκλογές. Όπως είπε και ο Μιχαήλ Γκάλες έκαναν πολύ καλή δουλειά. Οι εκλογές οργανώ, είχαν οργανωθεί καλά, χωρίς οργανωτικά προβλήματα δηλαδή και μπορούμε να το θεωρήσουμε θετικό αυτό. Και το 11 ήταν καλά τα πράγματα. Και η, το, και η τοτινή αποστολή μας είχε πει ότι όλα είχαν γίνει όπως έπρεπε. Χωρίς ιδιαίτερα οργανωτικά προβλήματα. Τώρα, όπως είπαν οι συνάδελφοι βέβαια, οι βουλευτικές εκλογές είναι το πρώτο η πρώτη φάση θα υπάρξουν μετά τον ίδιο μήνα προεδρικές και ίσως και δεύτερος γύρος των, τα Χριστούγεννα. Θα δούμε λοιπόν πώς μετά τις προεδρικές εκλογές θα διαμορφωθεί η πλειοψηφία. Παλιότερα η πλειοψηφία ήταν η Εναχντά που είχε πολύ μεγάλα ποσοστά και είχε αποφασίσει να συνταχθεί με δύο άλλα μικρότερα κόμματα που τώρα πια έχουν διαλυθεί. Αντίθετα υπάρχει μια επανεξισορρόπηση, μια νέα ισορροπία μεταξύ του Νίντα ΛΕΣ και της Εναχντά. Αυτό είναι κάτι καινούριο. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει, ποια πλειοψηφία θα διαμορφωθεί, εφόσον μάλιστα μπορεί η του ΝΕΣ να κερδίσει και τις προεδρικές. Μπορεί λέω. Γιατί το άλλο σημαντικό γεγονός είναι η αύξηση των εκλογέων. Πέρα από το γεγονός του διπολισμού, 90 του ΝΕΣ και ένα ΧΝΑΠ, υπήρχε και πολύ μεγάλος κατακαιρματισμό 1300 ψηφοδέλτια κάποια στιγμή. Πολύ δυσκολότερο ήταν λοιπόν να σηματιστεί κάποια πλειοψηφία. Μετά τις εκλογές του 11 λοιπόν το θέμα ήταν μπορούμε να δεχτούμε ότι υπάρχει κάποιο μετριοπαθές Ισλάμ στην εξουσία. Σήμερα το θέμα είναι ποια πλειοψηφία θα διαμορφωθεί μετά από την εμφάνιση του Νίντα Τουνές που είναι συνασπισμός βέβαια και με κοσμική βάση. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε μετά τις προεδρικές εκλογές. Εκεί θα δούμε πιο καθαρά αν η Εναχντά θα μείνει στην αντιπολίτευση ή στην εξουσία. Αν θα γίνει κάποιος νέος συνασπισμός ας πούμε, της Εναχντά με μικρότερα κόμματα για να υπάρξει κάποια άλλη ισορροπία. Ή αν θα αλλάξει η εξουσία και η πλειοψηφία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θέλω να συγχαρώ τους συναδέλφους οι οποίοι πήραν μέρος στην αντιπροσωπεία αυτή. Έγινε μεγάλη προσπάθεια και πράγματι με χαρά διαπιστώνουμε τις αλλαγές που έγιναν σε αυτή τη χώρα. Είναι ενθαρρυντικό που όλα τα κόμματα αποδέχθηκαν τα αποτελέσματα της διαδικασίας. Αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα. Ε, κάτι άλλο το οποίο βρίσκω θετικό. Τα λεγόμενα Ισλαμικά κόμματα βλέπω ότι αντιμετωπίζουν την κατάσταση στην Τινησία με έναν τρόπο ο οποίος ίσως να φανεί χρήσιμος και για άλλα Ισλαμικά κόμματα στη Μέση Ανατολή εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση και γι' αυτό είναι ένα παράδειγμα, ένα παράδειγμα το τινησιακό το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει έτσι ώστε και τα Ισλαμικά κόμματα να βοηθήσουν στην αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών. Ακούσαμε διάφορα για τους νέους οι οποίοι δεν πήραν μέρος τόσο στις εκλογές αυτές και αυτοί αποτελούν το μέλλον μας. Ε, για τις γυναίκες. Τι ακριβώς συνέβη, ποια ήταν η συμμετοχή των γυναικών. Κατανοούμε βέβαια ότι οι εκλογές είναι σημαντικό πράγμα, αλλά η δημοκρατία δεν είναι μόνο εκλογές. Ε, τι γίνεται με τους δημοκρατικούς θεσμούς στη χώρα αυτή. Εγώ είμαι νέος εδώ και θα με βοηθήσετε να καταλάβω τι βοήθεια απαιτείται στη συγκεκριμένη περίπτωση πέρα από τα εκλογικά θέματα έτσι ώστε να αποκτήσουν βαθιές ρίζες τα όργανα, τα θεσμικά, στην κοινωνία και στη Μέση Ανατολή γενικότερα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μποστινάρου, τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συνάδελφοι, θα είμαι σύντομος. Shows that they are continuously making... Η Ισία διαφοροποιείται για μια ακόμη φορά. Είναι μια χώρα η οποία μετά την Επανάσταση είναι σταθερή, είναι χώρα η οποία δεν έχει πάρα πολύ σημαντικές ριζοσπαστικές Ισλαμικές ομάδες. Είναι σαφές επίσης ότι οι εκλογές εξελίχθηκαν μέσα σε ειρηνική ατμόσφαιρα, καμία σύγκριση δηλαδή με άλλες αντίστοιχες διαδικασίες στην περιοχή του Μαγκρέμπ. Ε, δεν θέλουμε να δίνουμε μαθήματα σε κανέναν και ιδιαίτερα στις χώρες της περιοχής αλλά να δούμε ότι η Τινησία πήγε εντυπωσιακά καλά λαμβανομένων υπόψη των εντασσεών τις οποίες υφίσταται η χώρα αυτή. Ε, ταυτόχρονα η σχέση ανάμεσα στην Τινησία και την Ένωση είναι θεμελιώδης είναι η ανταπόκρισή μας σε μια έκκληση από πλευράς της ε, την πλευράς να στηρίξουμε την δημοκρατική διαδικασία. Αλλά και εμείς χρειαζόμαστε την Τινησία για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την δημοκρατική μας παρουσία στις χώρες ε, του Μαγκρέμπ. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με το Μαρόκο, την Αλγερία και την Τινησία αλλά μόνο εφόσον το ζητούν μπορούμε να βοηθήσουμε και έτσι θα επηρεάσουμε και θετικά εξελίξεις στις υπόλοιπες χώρες. Πρέπει να ακούσουμε το τι θέλουν οι μετριοπαθείς Ισλαμικές δυνάμεις έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση η οποία οδήγησε στις εκρήξεις ε, σε όλες τις χώρες της περιοχής. Έχει επίσης ε, ε, να δούμε τι γίνεται με με τα χρήματα του Μπεναλή τα οποία έχουν παρακρατηθεί σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην δίνουμε μόνο μαθήματα, να αντιμετωπίσουμε αυτήν την δραματική πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αντιμετωπίσει δίκαια τα ποσά αυτά που έχει κλέψει ο Μπεναλή. Ε, και στην Ευρώπη και στη Σαουδική Αραβία βέβαια που υπάρχουν αντίστοιχα αντίστοιχα πως Τώρα, για το Euromed, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, το Euromed θα πρέπει να παίξει έναν πιο σημαντικό ρόλο, εργαζόμενο για την σταθεροποίηση της περιοχής στο μέλλον και για την έβρεση τρόπων περαιτέρω σταθεροποίησης των χωρών οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικά θέματα όπως η Λιβύη. Ε, χώρες οι οποίες χρειάζονται την συνεργασία μας και την συνεργασία της Τινησίας φυσικά. Μιλάμε για μια ομάδα χωρών η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα. Πάντως συγχαίρω τους Τινήσιους γιατί πραγματικά ξεπέρασαν αυτό το εμπόδιο με επιτυχία και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί τους έτσι ώστε να μάθουμε και από αυτούς το τι πρέπει να γίνεται στο μέλλον. Ευχαριστώ. Και εγώ θα, θα Ήθελα να δώσω εν τέλει το λόγο στον κύριο Γκάλε. Σα. ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Απλώ για να κλείσω τη συζήτηση και να απαντήσω σε ορισμένα από τα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν πρώτα απ' όλα για την συνεχιζόμενη συνεργασία. Νομίζω ότι υπάρχει ευρεία συνένεση ότι πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, ότι εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εμπλακούμε. Έχουμε προσπαθήσει μέσα από την UNDP, τον Οργανισμό ανάπτυξη του Ηνωμένου, των Ηνωμένων Εθνών, να έλθουν να συμμετάσχουν και αυτοί σε μια συνδιάσκεψη που θα γίνει στην Ισία για την οργάνωση πολιτικών ομάδων. Μας έχουν ε, ζητήσει και εμείς να συμμετάσχουμε και να δώσουμε τη δική μας ε, άποψη για το πώς πρέπει να οργανωθούν οι πολιτικές ομάδες, πώς γίνονται οι πολιτικοί συνασπισμοί. Όλα αυτά θα τους ενδιαφέρουν να τα γνωρίζουν και από την ευρωπαϊκή πλευρά. Όλα αυτά λοιπόν επίκυνται από τις αρχές του 2015 σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των γυναικών από την, Επιτροπή, από την Εκλογική Επιτροπή μας είπαν ότι ήταν περισσότερες γυναίκες οι οποίες καταγράφηκαν στα εκλογικά μητρό από τους άνδρες και μέσα στην κοινωνία των γυναικών, των πολιτών με υπήρξε έντονη συμμετοχή των γυναικών γιατί φυσικά είχαν πολύ περισσότερα να χάσουν αν το Σύνταγμα πήγαινε προς τη διατεύθυνση της Ισαρίας. Υπήρξε λοιπόν μεγάλη συμμετοχή των γυναικών και των οργανώσεων των γυναικών. Την ίδια τη μέρα των εκλογών δεν έχω τώρα την εντύπωση ότι υπήρξε μια ε, καταμέτρηση χωριστά των ανδρικών και γυναικείων ψήφων. Δεν ξέρω ακριβώς πώς ήταν η συμμετοχή τους, αλλά είδα μεγάλες ουρές στα εκλογικά τμήματα που ήταν μικτές, δεν ήταν μόνο άντρες ή μόνο γυναίκες. Αυτό το οποίο είναι και ενδιαφέρον σε σχέση με τους εκλογικούς καταλόγους και τα ψηφοδέλτια, υπήρχε πάντα η υποχρέωση να είναι εναλλάξ τα ονόματα ανδρών και γυναικών και συμμετοχή γυναικών σε επίπεδο 50%. Το εκλογικό σύστημα τώρα, την τελευταία φορά που είχαμε μονάχα ένα μεγάλο κόμμα, είχε οδηγήσει στο να λειτουργεί το αναλογικό σύστημα στις περιφέρειες που είχαμε maximum 10 εδρών. Όταν έχει όμως κανείς ένα μεγάλο μονάχα κόμμα, όπως την προηγούμενη φορά, και έχοντας πάντα τις περισσότερες φορές άνδρες ως νούμερο ένα στον κατάλογο, ε, το αποτέλεσμα ήταν ότι μόνο το μεγάλο κόμμα, το ενάχτα, είχε αρκετές γυναίκες που εξελέξαν τώρα, επειδή έχουμε περισσότερες γυναίκες, δεν ξέρω ακριβώς πόσες, έχουμε πολλές περισσότερες γυναίκες και προέρχονται από τα δύο κύρια κόμματα. Ήταν οι περισσότερες περιπτώσεις οι άνδρες οι οποίοι ήταν επικεφαλής των ψηφοδελτίων και το γεγονός ότι υπήρξε κομματισμό όπου τουλάχιστον το δεύτερο άτομο σε κάθε ε, ψηφοδέλτιο εξελέγει είχε περισσότερες γυναίκες. Ε, έχουμε έτσι λοιπόν την πιθανότητα να έχουμε περισσότερες γυναίκες εν τέλει. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Προεδρεύων. Σίγουρα θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό και πρέπει το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει υποστήριξη στη σταθερότητα της ε, Βόρειας Αφρικής. Ερχόμαστε τώρα σε ένα άλλο σημείο. Το πρωτόκολλο λοιπόν για τη Μεσογειακή Συμφωνία, ε, για το σύμφωνο μάλλον της Μεσογειακής Συνεργασίας σχετικά με την Τινησία. Από τον Νοέμβριο λοιπόν, αρχές μάλλον Νοεμβρίου αυτού του μήνα, ε, υπάρχει το θέμα της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας με την Τινησία για την ε, λήψη υπόψη προσχώρηση των τελευταίων δύο χωρών. Πάρα πολύ σύντομα λέει ο κ. Παντσέρη, πρόκειται για μια δικασία τεχνική η οποία λαμβάνει υπόψη την είσοδο της Βουλγαρίας και της Ρωμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 2007 επηρεάζεται νομικά θα έλεγα η συμφωνία την οποία έχουμε με τις δύο αυτές χώρες. Άρθρο 217, 218, ε, α, β και γ τις συνθήκες. Τίποτα αντιρρήσεις δεν υπάρχουν, είναι τεχνικό το θέμα για την εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλου συνεργασίας και στις δύο νέες εισαγωγικά χώρες. Λοιπόν, να θυμηθούμε το χρονοδιάγραμμα. Θα ψηφίσουμε την 1η Δεκεμβρίου του 2014 στην Επιτροπή και θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια τον Ιανουάριο του 2015. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Ο πρεσβευτής τη Νησία θέλει να πει κάτι ακόμα. Απλώ να σα δώσω μια διευκρίνηση για τι 217 έδρε εξελέγησαν 68 γυναίκε, 31% λοιπόν των εκλεγμένων στην Τινησία είναι στο Τινησιακό Κοινοβούλιο οι γυναίκες. Αυτά. Στη Σας ευχαριστώ. Εάν δεν υπάρξει κάτι άλλο που θέλετε να πείτε, μπορούμε να κλείσουμε τη συνεδρία σε αυτή. Τρισήμιση το απόγευμα σε μια άλλη αίθουσα συνεχίζουμε. Ευχαριστώ.